Ε. So, going to start and resume. The first point for, for this morning, this afternoon, sorry. Καλησπέρα σας. Ξεκινάμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Έχουμε κοινή συζήτηση. Αχ, χρειάζομαι περισσότερο καφέ. Έχουμε λοιπόν κοινή συζήτηση για την απαλλαγή σημεία 23 μέχρι και 28 στην ημεριασία διάταξη. Ε, είμαστε εδώ εγώ και ο εισηγητής. Αυτός είναι ο εισηγητής. Δηλαδή εγώ. Και πρέπει λοιπόν να <laughs> δώσουμε την ε, γνωμοδότησή μας για την απαλλαγή της DG Κλίμα, DG Περιβάλλον, DG 5 τέλος πάντων γενικές διευθύνσεις, ΕΜΑ, ΕΚΑ και ΕΦΣΑ. Βεβαίω πρόκειται για το, την χρήση 2018, διότι οι απαλλαγέ γίνονται πάντοτε δύο χρόνια μετά και θα ήθελα να αναφέρω κάποια σημεία που θεωρώ ότι είναι σημαντικά. Ε, το πρώτο είναι βεβαίως να υπογραμμίσω ότι το ελεγκτικό συνέδριο ε, ε, ενέκρινε τους λογαριασμούς 2018 όλων των οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι δηλαδή οι λογαριασμοί ήταν αξιόπιστοι και αφυσικά είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Να πούμε επίσης ότι οι οργανισμοί εργάζονται, συνεργάζονται περισσότερο μεταξύ τους, είναι πιο συνεπείς άρα και ε, κάνουν οικονομίες έτσι στη χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Και αυτό αποδίδει καρπούς. Η ΕΜΑ, η ΕΦΣΑ και η ΣΥΤΙΣΗ έχουν εργαστεί, συνεργαστεί για την αντίσταση για τα, στα αντιβιωτικά και άλλοι οργανισμοί έχουν δουλέψει από κοινού για τα πειράματα σε ζώα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζουμε όταν πρόκειται για οργανισμούς και υπηρεσίες ότι ενώ τα αιτήματα είναι ε, αυξανόμενα, ο προπολογισμό δεν ακολουθεί πάντοτε και γι' αυτό μας ε, χρειάστηκε να μειώσουν κάποιες δραστηριότητες γιατί δεν είχαν αρκετούς πόρους, πράγμα το οποίο είναι εν γέννη αντιφατικό με την εντολή που εμείς τους δίναμε, τις δικές μας δηλαδή απαιτήσει. Πρέπει λοιπόν να υπογραμμίσουμε την ανάγκη να έχουμε και τα κατάλληλα κονδύλια πράγμα που κάνουμε και ευτυχώς ε, κερδίζουμε το ημάχη αυτή στον προπολογισμό για το 2020. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε την απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς για το 2018. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή, θα ήθελα να ε, μιλήσω πιο συγκεκριμένα για την ΕΝΤΕΤΖΕ κλίμα στη Γενική Διεύθυνση για το Κλίμα και να υπογραμμίσω ένα σημείο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό και επί του οποίου θα ακούσουμε και την Γενική Διεύθυνση Κλίμα, ε, δηλαδή του σημαντικού κινδύνους όσον αφορά την ασφάλεια των ε, συστημάτων ETS, γιατί αυτό το αποθεματικό υπάρχει από το 2010 και έχουν γίνει απόπειρε για επίλυση του προβλήματος ε, πληροφορικής και ασφάλειας αυτού του, αυτής της αγοράς, αλλά όχι ικανοποιητικά φτάσαμε σε κάποια φάση να έχουμε προτάσεις για το Green Deal, το πράσινο σύμφωνο. Σίγουρα θα μας δώσει κάποιους δρόμους για μεταρρύθμιση της αγοράς του άνθρακα που ε, θα την καταστήσει πιο σημαντική για την ε, ευρωπαϊκή πολιτική κλίματος. Δεν μπορούμε να διακινδυνεύσουμε μια τόσο σημαντική αγορά να υπόκειται σε ανασφάλεια πληροφορική. Είναι απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Και άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό η Γενική Διεύθυνση Κλίμα να επανέλθει με συγκεκριμένες προτάσεις. Το άλλο στοιχείο που δεν μας ικανοποιεί έχει να κάνει με την αναφορά του αυτό που ονομάζουμε Climate Instrument, ε, μέσο για το κλίμα. Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον ε, γιατί στο παρελθόν δεν μπορούμε να αλλάξουμε τίποτα, αλλά στο μέλλον αντιθέτως μπορούμε. Δηλαδή, οι γραμμές αναφοράς για το climate mainstreaming να είναι αρκετά συγκεκριμένες ώστε να μπορούμε να δούμε ακριβώς τι αλλάζει και τι παραμένει το ίδιο. Σήμερα αυτό δεν ισχύει. Θα δουλέψουμε από αυτού από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή Προπολογισμού και εκεί μια από τις δεσμεύσεις που θα πρέπει να αναλάβουμε στο πλαίσιο του Green Deal είναι να ενισχύσουμε την ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού του συνόλου του PDP και αυτό που ονομάζουμε Green Budget budgeting, δηλαδή πράσινος προϋπολογισμός, ε, θα πρέπει να γίνει για, ολόκληρες, για όλες μάλλον τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει λοιπόν για όλα αυτά τα ποικίλα θέματα να μπορούμε να δούμε με λεπτομέρειες ε, ακριβώς που ε, γίνεται η ευθυγράμμιση, η πράσινη ευθυγράμμιση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας παρέχει τα έγγραφα όχι μόνο η ΕΝΒΗ αλλά και του προπολογισμού, του ελέγχου προπολογισμού, όλες οι αρμόδιες επιτροπές δηλαδή να μπορούν να αξιολογήσουν την ευθυγράμμιση με τη Συμφωνία του Παρισιού. Αυτό ισχύει για το κλίμα αλλά και για τη βιοπικιλότητα, πράγμα που συζητήσαμε με την ΕΤΕΠ πριν από λίγο και τις ψηφοφορίες που κάναμε σήμερα το πρωί. Δύο σημαντικά λοιπόν σημεία ε, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με μια αγορά άνθρακα που δεν είναι ασφαλής όσον αφορά την πληροφορική και ένα θέμα σημαντικό είναι το πρασίνισμα ε, όλων των πολιτικών. Αυτά τα δύο σημεία ήθελα να τονίσω που είναι στρατηγική σημασία κατά τη γνώμη μου. Θα δώσω τώρα το λόγο στους διάφορους κοιόδης για αυτό το θέμα και θα ξεκινήσω από τον Στανισλάβ Πολζάκ από το ΕΛΚΑ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά εγώ υποστηρίζω την απαλλαγή τόσο για την Κομισιόν στο πλαίσιο της, ε, των όσων προβλέπονται από την ημερήσια μας διάταξη για την οικονομική χρήση 2018, καθώς επίσης και για τις πέντε αποκεντρωμένες ε, πέντε αποκεντρωμένους οργανισμούς. Μπορούμε να πούμε πως εν γέννη είμαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που χρησιμοποίησε τα κονδύλια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωστόσο υπάρχει πάντοτε και ένα περιθώριο λιγμού, ένα περιθώριο βελτίωσης και θα ήθελα να παραθέσω κάποια συγκεκριμένα σημεία. Όσον αφορά την Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ, να υπογραμμίσω ότι κυρίως στο πρόγραμμα LIFE υπήρχαν αρκετές, αρκετά σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών που ήταν δύο φορές μεγαλύτερες από αυτές του 2017. Επίσης, σε σχέση με το πρόγραμμα Life πάντοτε, θα πρέπει να πούμε πως η κατάσταση είναι κάπως τεταμένη, γιατί από ό,τι φαίνεται η Γενική Διεύθυνση θα πρέπει να ξαναδεί την οργάνωσή της και να υιοθετήσει σημαντικές συστάσεις για να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Όσον αφορά την γάμα δέλτα κλίμα, την αναφέρατε και συμφωνώ με τα όσα είπατε. Ε, να επιτρέ... επιτρέψατε μου να πω δύο λόγια για τη Γενική Διεύθυνση Σαντέ Υγεία. Εδώ θα πρέπει να δούμε ότι το ποσοστό σφάλματος ε, στις δραστηριότητες αυτής της Γενικής Διεύθυνσης δεν ξεπερνά το κατόφλι του 2%. Δεν είναι δηλαδή πολύ σημαντικό ποσοστό. Το ελεγκτικό συνέδριο δε ε, έχει διαπιστώσει ότι πάνω από το 98% η εκτέλεση ήταν σωστή. Ωστόσο, αρκετές ε, πληρωμές δεν μπόρεσαν να γίνουν εγκαίρως από την Γενική Διεύθυνση Υγεία και αυτό θα πρέπει να βελτιωθεί λοιπόν και να προχωρήσω τώρα σε κάποιες ε, παρατηρήσεις όσον αφορά τις δραστηριότητε των οργανισμών που είναι επίσης ε, τμήμα αυτής της κοινή συζήτηση. Όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Περιβάλλον, θα ήθελα να πω να υπογραμμίσω πως αυτός ο οργανισμός παίζει πανευρωπαϊκό ρόλο, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός διότι αφορά και τη συνεργασία με τρίτες χώρες εκτός Ένωσης. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού του οργανισμού διαπίστωσε ότι ο οργανισμός αντιμετωπίζει έλλειψη ε, κονδυλίων, όπως και εσείς υπογραμμίσατε κύριε Πρόεδρε, και ε, Άρα περιορίζονται οι δυνατότητες αντίδρασης και δράσης σε σχέση με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι η δική μας ε, κοινοβουλευτική δραστηριότητα θα πρέπει να προσανατολιστεί προς την στήριξη της αύξησης των πόρων για αυτόν τον οργανισμό. Είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο για όλους τους οργανισμούς, ε, γιατί ε, αποδίδουμε, μάλλον αναθέτουμε όλο ένα και περισσότερα καθήκοντα και αποστολές σε αυτούς τους οργανισμούς, ωστόσο τα χρήματα παραμένουν στο ίδιο επίπεδο. για τον οργανισμό για την υγεία. Για ε, τα φάρμακα, μας συγχωρείτε. Εδώ ε, θα μετακινηθεί ο οργανισμός αυτός από το Λονδίνο στο Άμστερνταμ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό για το 2018 και αυτό επηρέασε βεβαίω και τι δραστηριότητε του οργανισμού η μετακίνηση. Όμω, κατά τη γνώμη μου, καταφέραμε να διαχειριστούμε <coughs> την μετακίνηση, ακόμα και αν κάποιε θέσει ε, δεν έχουν ακόμα καλυφθεί. Ορισμένοι εργαζόμενοι δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις τους, οπότε υπάρχει κάποια έλλειξη προσωπικού. Γιατί οι οργανισμοί πρέπει να αντιμετωπίσουν και εκείνοι τον αντίκτυπο του Brexit. Το βλέπουμε στην περίπτωση του οργανισμού για τα φάρμακα. Είναι σημαντικό να το υπογραμμίσουμε και ταυτόχρονα να τους καλέσουμε να τηρήσουν τις αξίες της ε, διαφάνειας ε, και θα προτείνω κάποιες ε, μικρές τροπολογίες. Αλλά όπως είπα και το επαναλαμβάνω κλείνοντας, ότι συμφωνώ απόλυτα με τη δική σας γνώμη Δηλαδή να χορηγήσουμε την απαλλαγή σε όλους τους οργανισμούς αλλά και στην Επιτροπή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές. Η κυρία Μπένοβα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω στα σλοβακικά. Όσον αφορά τους ε, αποκεντρωμένους αυτούς ε, οργανισμούς, ε, υπάρχουν επαρκές δραστηριότητες και υπήρξε σε όλες τις περιπτώσεις σωστή διαχείριση των κονδυλίων. Δεδομένου του φόρτου εργασίας που αυξάνεται στους οργανισμούς αυτούς, ετησίως ε, ε, αυξάνεται ε, η δουλειά που έχουν να κάνουν χωρίς αύξηση του προϋπολογισμού. Γι' αυτό προτείναμε να δοθούν επαρκή κονδύλια για να καλύψουν όλες τις δραστηριότητε. Όσον αφορά τους οργανισμούς αυτούς, θα πρέπει να εστιαστούμε για την προστιθέμενη αξία που προσφέρουν αυτοί οι οργανισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά και στη βοήθεια που παρέχουν στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Όλοι οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί παίζουν σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δουλειά τους πρέπει να επικοινωνείται με επαρκή τρόπο και το 2018 παρατηρήσαμε ότι ε, έχουν και μεγαλύτερη προβολή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ε, και στα μέσα γενικότερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η διαφάνεια είναι μια από τις ε, αρχές κλειδί που πρέπει να διέπει τη δραστηριότητα των οργανισμών αυτών. Αφού δεν υπήρξαν κάποια προβλήματα, εμείς συνεχίζουμε με την ίδια αρχή διαφάνειας. Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και να ε, πω ότι σε, όλες τις, ε, σε όλους τους οργανισμούς υπήρξε ισότητα ε, φίλων. Σε κάποιους οργανισμούς υπάρχουν και περισσότερες γυναίκες από άντρες, οπότε αφού μιλάμε για ισότητα μεταξύ των φύλων, θα πρέπει να αναρωτηθούμε αν υπάρχουν αρκετοί άντρε τελικά σε αυτού του οργανισμού. Ε, το, η ομάδα μα θα κάνει διάφορε προτάσει. Και είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που για το 2020 λήφθηκε υπόψη μία από τις δικές μου προτάσεις όσον αφορά τη μεταβολή πόρων για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος ύψους 1,3 εκατομμυρίων, κάτι που επέτρεψε να αυξηθούν οι πόροι που έχει ο οργανισμός. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στους άλλους οργανισμούς. Αλλά βάσει των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας, μπορούμε να χορηγήσουμε την απαλλαγή στην ε, Επιτροπή όσον αφορά τους ε, πόρους για τους οργανισμούς αυτούς ε, για το έτος 2020 καθώς και στην στο πλαίσιο της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτός μικρόφωνου. Για τους πρασίνους, η κυρία Γιούτα Παύλος. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, ευχαριστούμε για το σχέδιο γνωμοδότησης. Πολλοί από τους συναδελφούς μου το είπαν ήδη ότι η απαλλαγή θα πρέπει φυσικά να βοηθηθεί αφού έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά αυτοί οι οργανισμοί και οι Κομισιόν και εδώ δεν σπαταλώνται τσάμπα τα χρήματα των φορολογουμένων. Εμεί έχουμε υποβάλει κάποιε τροπολογίε και θα σα θίξω κάποια ζητήματα τώρα για την Επιτροπή. Ο στόχο του 20% ένταξη του κλίματο ε, ε, σε όλε τι πολιτικέ ε, δεν επετεύχθη αυτή τη φορά. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε για να επιτευχθεί αυτό ο στόχο. Ειδικότερα επειδή θέλουμε να αυξήσουμε και το στόχο μάλιστα για να καλύψουμε τις ε, προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Οπότε ελπίζω να υπάρξει κάποια στρατηγική από την Κομισιόν ώστε να διασφαλιστεί η εκπληρώση του στόχου. Θα ήθελα να δούμε τους αντίστοιχους οργανισμούς. Ε, είχαμε τον κύριο Χάνσεν από την ΕΚΑ εδώ χθε. Αυτός μας έδωσε ε, μια πολύ καλή εικόνα για το ποια είναι τα καθήκοντα του οργανισμού. Μας μίλησε για αύξηση των ελέγχων που πρέπει να πραγματοποιούν. Νομίζω ότι η ΕΚΑ αναλαμβάνει τεράστιε ευθύνε για την ασφάλεια τόσο των εργαζομένων όσο και των καταναλωτών και αντιμετωπίζουν δύσκολες έπογες ε, ε, χρηματοδοτούνται μέσω τελών. Αλλά ποτέ δεν ξέρει κανεί πόσα τέλη τελικά θα εισπράξει μέχρι το τέλο του έτου. Οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο ο σχεδιασμό ε, των ανθρώπινων πόρων. Ανάλογα με τι ανάγκε. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, θα έπρεπε να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κατά πόσο θα μπορούσε να υπάρχει ένας καθορισμένος προϋπολογισμός για την ΕΚΑ και τα τέλη να ε, καταλήγουν στο γενικότερο προπολογισμό τη Ένωση. Αυτό θα έκανε τον προγραμματισμό πολύ ευκολότερο. Επίση, πιστεύω ότι ε, ετούντες που ε, αποπειρώνται απάτη ή που δεν συμμορφώνονται θα πρέπει να πληρώνουν μεγαλύτερη συνεισφορά γιατί αυτή είναι που δυσκολεύει την κατάσταση αν οι φάκελοι ολονών ήταν εντάξει δεν θα ήταν ε, τόση πολλή δουλειά για τον οργανισμό να ψάξει να βρει τα παραθυράκια. Ε, όσον αφορά την ΕΦΣΑ, ε, σε συζητήσει που είχαμε ψηφοφόρου, πολλοί κόσμοι ενισχύει για την ασφάλεια των τροφίμων. Η ΕΦΣΑ, λοιπόν, θεωρώ ότι έχει τεράστιε ευθύνε να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που βάζουμε στο πιάτο μα είναι ασφαλή. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να, να οι αξιολογήσει να γίνονται ανεξάρτητα και αναφέρθηκε ότι η διετής περίοδος όντως εφαρμόζεται αλλά όχι πάντα στην πραγματικότητα γιατί υπάρχει το ε, οικονομικό όριο του 25% Οπότε δεν υπάρχει πλήρης απορρόφηση όταν λοιπόν ε, η χρηματοδότηση γίνεται από τη βιομηχανία ε, σε κάτω από 25% θεωρεί ανεξάρτητο συμπρογνώμων. Δεν μπορεί να γίνεται αυτό, διότι στην ομάδα για την εξέταση των γονιδίων το 50% των εμπειρογνωμόνων ε, που γνωμοδοτούν είχαν οικονομικούς δεσμούς με εταιρείε που εργάζονται ε, σε γονιδιακές θεραπείες και σε σχετικά φάρμακα. Οπότε δεν επαρκώς ανεξάρτητοι ώστε να γίνεται πραγματικά σωστή αξιολόγηση των κινδυνών για τους χρήστες και το περιβάλλον όταν έχεις ανθρώπους εκεί οι οποίοι έχουν οικονομικούς δεσμούς με τους παραγωγούς. Όσον αφορά την αίμα, τα συλληπιτριά μου, αυτοί πραγματικά υπέστησαν όλο το άχθος του Brexit όπως αναφέρθηκε ήδη ε, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που τους αναμένει. Έχουν να, ε, να απέναντί τους ε, εταιρείε με μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο. Έχουν να δημοσιευτούν κλινικά δεδομένα εδώ και πάνω από ένα χρόνο, διότι οι φαρμακευτικές εταιρείε λένε είναι ιδιωτικά. Δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε διαφανείς, οπότε ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων πρέπει πάντα να πηγαίνει στα δικαστήρια και να μάχεται. Οπότε χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ECDC, και εκεί ανησυχώ λίγο. Θεωρώ ότι ε, για το 96% των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχουν υποβληθεί οι δηλώσει σε εγκρούσει συμφερόντων. Δεν καταλαβαίνω γιατί είναι τόσο δύσκολο. Θα πρέπει να εφαρμοστεί και για την EEA, την, που μείνει ιδιαίτερα προσφυλή, γιατί εγώ είμαι το άτομο επαφής ε, να πω εδώ ότι η ΕΕ είναι αρμόδια για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης ε, βοηθώντας να επιτυγχάνονται σημαντικές και μετρήσιμες πρόοδοι ε, στο περιβάλλον στην Ευρώπη. Έχουν διάφορα δεδομένα, διάφορες, διάφορες πληροφορίες σε αυτόν τον οργανισμό, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος Ε, για να βρει κανεί όμω τι να κάνει πρέπει να ψάχνει μέσα στην ιστοσελίδα του δυο τρει μέρε. Και όπω είπα, τα καθήκοντά του για να συλλέγουν τα δεδομένα, να τα αξιολογούν, να διαπιστώνουν ε, ποια είναι η κατάσταση του περιβάλλοντο, δεν θα πάψουν. Αντιθέτω, θα είναι περισσότερα αυτά τα καθήκοντα, γιατί θα παίξουν πολύ σημαντικότερο ρόλο από ό,τι στην προηγούμενη θητεία. Γι' αυτό χρειάζονται βιώσιμη χρηματοδότηση, όχι μόνο στο 2020, αλλά και στο επόμενο πολιτέ μεσονομικό πλαίσιο. Και ο διευθυντή μου είπε ότι του έχουν ήδη πει ότι θα πρέπει να αναμένει περικοπές στον προϋπολογισμό προσωπικού. Δεν καταλαβαίνω πώς θα καταφέρουν να κάνουν τη δουλειά τους όπως χρειάζεται, αν έχουν λιγότερους ανθρώπους και περισσότερα καθήκοντα. Ελπίζω λοιπόν όλα τα μέλη εδώ της Επιτροπής να απαιτήσουν ένα βιώσιμο προπολογισμό για αυτόν τον οργανισμό. Προσβλέπω να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε ε, για τις τροπολογίες και την τελική γνωμοδότηση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Any other speaker? No. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος ομιλητής, η Κομισιόν θέλει να πάρει το λόγο. Τυχαία. Ας ξεκινήσουμε με την DG Κλίμα, Ένδη και μετά Σάντε. Thank you, Mr. Chairman. Um, Rudy van Orenbeek uh, from DG Climate Action on behalf of the Commission. Θα ήθελα εκ μέρους της Επιτροπής να πω τα εξής. Πρώτα απ' όλα, χαιρετίζουμε την πρότασή σας για την χορήγηση τις ε, απαραγές. Όσο για τα θέματα που θέσατε στην ΙΤΕΣ, βεβαίως όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για τον ε, ακνογωνιαίο λίθο του οικίματος. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, τα ε, δισεκατομμύρια ευρώ. Ξέρουμε ότι πριν από χρόνια ήταν πολύ λιγότερα κατά 5%. Βλέπουμε λοιπόν πόσο αναπτύσσεται ο τομέα αυτέ. Σαν το χρηματιστήριο, είναι πολύ πλοκό το σύστημα για να το χειριστεί κανεί. Και μπορώ να σα πω πολλά πράγματα γιατί πώ μπορέσαμε να το διαχειριστούμε και να το βελτιώσουμε σε καθημερινή ή σε αιτήσια βάση. Έγινε ε, εσωτερικός ε, οικονομικός έλεγχος, ε, κάναμε καλό σχεδιασμό, ανάλυση του ρίσκου. Το 2018 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με τα τελευταία στάνταρ, το συμπέρασμα μας είναι ότι δυστυχώς το σύστημα ακόμη δεν είναι σε επίπεδο να αποκρίνεται σε όλα τα στους κανόνες ασφαλείας. Αυτό το οποίο όμως ε, κατορθώσαμε να κάνουμε είναι να μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας και ποιότητας στο Λουξεμβούργο, το hardware, αλλά υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, συνθήκες τις ε, δύσκολες και με την Γενική διάθεση Digit και με άλλες γενικές διευθύνσεις, δεδομένου ότι το όλο σύστημα και τα μέσα που χρησιμοποιούν είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ε, ε, Επιτροπή. Μιλούμε για πόρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση και για χρήματα τα οποία θα μπορέσουμε να δούμε για να κάνουμε και νέες επενδύσεις στον τομέα το προτεθείς περιβάλλοντος και βεβαίως πρέπει να πω ότι για να μην επαναλάβουμε τις... τα προβλήματα του παρελθόντος για την ε, όλη διακυβέρνηση προσπαθούμε να βρούμε νέες εναλλακτικές λύσεις. Δεν ξέρουμε αν θα πρέπει στην έκθεση για το 2019 τι επιφυλάξει που έχουμε, αν πρέπει να τι άρουμε ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να σα αποκαλύψω τίποτα περισσότερο. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και δεδομένου ότι πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, θα σα ενημερώσουμε έγκαιρα. Τώρα, όσον αφορά την, ε, το mainstreaming, τον ορθολογισμό σε θέματα κλίματος. Πρέπει να πω ότι με διάφορες τροπολογίες προστίθονται 10 εκατομμύρια ευρώ για το 2020. Αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μας. Θα τα χρησιμοποιήσουμε για θέματα προστασίας ε, και για το πρασίνισμα που είναι το κέντρο της πολιτικής της Κομισιόν πάρα πολύ προσεκτικά αυτά τα κονδύλια. Επίσης, για το παρόν δημοσιονομιστικό πλαίσιο ε, ο στόχος μας έχει επιτευχθεί κατά 99,3%. Πρόκειται για μία δραστηριότητα η οποία δεν έχει 100% επιτυχία γιατί ήταν και πρωτοκόρ, πρόρος ή άλλως. Εν πάση περιπτώσει και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε στο 25%. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσουμε να θεσπίσουμε πιο αυστηρά μέτρα αναφοράς και εποπτείας με εκπλήσει το ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας ε, πίνακας εμπεριστατωμένος ώστε να μπορέσουμε να, σας, να έχουμε και να, πάρουμε πληροφορίες, να σας δώσουμε πληροφορίες για τη λεπτομερή κονδύλια τα οποία έχουν δοθεί σε κάθε δραστηριότητα. Αλλά θα έρθω σε επαφή με την Επιτροπή Προϋπολογισμών. Το Green Reporting Αυτά οι αναφοράς δηλαδή είναι κάτι το οποίο καλύπτει όλους τους τομείς. Ξεπερνάει τον τομέα της δικής σας ε, αρμοδιότητας. Θέλουμε λοιπόν συνεργασία με εσάς να μπορέσουμε να αναπτύξουμε αυτή τη νέα έννοια. Όλα αυτά βεβαίω την προστασία όλων την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα συνεχίσω χωρίς να καλύψω τα σημεία τα οποία ήδη κάλυψε για το κλίμα ο Ρούντι. Θα σταματήσω στο πρόγραμμα LIFE. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο, το οποίο από τις δικές μας γενικές διευθύνσεις και των δύο για βιώσιμα προγράμματα. Και Είπατε εσείς ότι έγιναν κάποιες ε, πληρωμές με καθυστέρηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί το πρόγραμμα. Σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιοι, υπήρχαν κάποια προβλήματα για κάποιους δικαιούχους οι οποίοι έλαβαν τα κονδύλια που τους αναλογούσαν αργότερα. Αν κάνει κανείς μια προσεκτική ανάλυση, θα δει ότι αυτές οι πληρωμές καθυστέρησαν για τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή με τα Life project βάσει των προηγούμενων κανονισμών. Τώρα αλλάζουμε και συγχρόνως το 2018 η Γενική Διεύθυνση ΕΝΒΗ ανέθεσε σε εξωτερικό προσωπικό σε μεγάλο βαθμό την υλοποίηση του προγράμματος LIFE. Όντως υπήρχε λοιπόν πρόβλημα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω όμως, δεδομένου ότι έχουμε ήδη τις στατιστικές για το 2019, ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και βρισκόμαστε τώρα στους κανονικούς μας ε, ε, ρυθμός, δηλαδή κάποιες μικροκαριθερήσεις 2-3%. Βεβαίως, με μεγάλη ταχύτητα λοιπόν μπορώ να επιβεβαιώσω ότι προχωρούμε, προσπαθούμε να κλείσουμε, να ολοκληρώσουμε όλες τις δράσεις και τα προγράμματα επιτόπου. Αυτή τη στιγμή μέσω της ΕΑΣ με θέτουμε σε εφαρμογή περισσότερα προγράμματα ευρύτερου περιεχομένου και με την ε, συμμετοχή πολλών χωρών. Θα ήθελα επίσης να χαιρετήσω τα σχόλια που κάνατε για την Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος. Ξέρουμε ότι είναι ένας οργανισμός που κάνει πολλά πράγματα και είναι κύριος πυλώνας των αναφορών σε θέματα περιβάλλοντος, κλίματος και βοηθάει και την Επιτροπή αλλά και εσάς ώστε να κάνει, να έχει μια σωστή κρίση για πάρα πολλές πολιτικές που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον. Άρα χαιρετίζουμε το γεγονό ότι αποφασίστηκε να δοθούν στον οργανισμό αυτό στο πλαίσιο του προπολογισμού του 2020 κάποια συμπληρωματικά κονδύλια και μπορώ να σας, να διασφαλίσω ότι θα χρησιμοποιηθούν πλήρως, πλήρως για το Green Deal. Και όχι μόνο εμείς, αλλά όλη η Επιτροπή προσπαθεί να έχει στο τομέα αυτό τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Καταλαβαίνουμε επίσης το πρόβλημα της ΕΚΑ που ανέφεραν οι συνάδελφοί σας για την μη βιωσιμότητα, έτσι δεδομένου ότι πρόκειται για ένα οργανισμό ο οποίος βασίζεται σε ε, συνδρομές Όσον αφορά λοιπόν τα δημοσιονομικά της, προσπαθούμε πολύ, κυρίως όταν ανατίθενται και νέα κατήθηκοντα στους οργανισμούς μας, προσπαθούμε, επαναλαμβάνω, να πείσουμε και τις άλλες υπηρεσίες, καθώς και το όλο σύστημα, ότι έχουμε οικονομικούς περιορισμούς, δεν μπορούμε να αυξήσουμε τους πόρους, δεν μπορούμε να αυξήσουμε το προσωπικό, αλλά προσπαθούμε με κάποιους άλλους τρόπους να δώσουμε συμπληρωματικά κονδύλια σε οργανισμούς όπως, όπως προανέφερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας Ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τα σχέδια γνωμοδότησης που προτείνουν την χορήγηση απαλλαγής για τις αποκεντρωμέ... τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Όσον αφορά τα προγράμματα υγείας και ασφάλειας των τροφίμων, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε κάνει ό,τι το δυνατό για να εφαρμόσουμε πλήρως τα προγράμματα ε, και όσον αφορά το σχόλιο που αφορά την καθυστέρηση καταβολής πληρωμών στο πρόγραμμα ασφάλειας των τροφίμων, λάβαμε τα απαραίτητα μέτρα στη διάρκεια του 19 ώστε τα μέτρα να μπουν και πάλι, μάλλον οι πληρωμές να μπουν και πάλι στη σωστή πορεία και να έχουμε καλά αποτελέσματα για το 2019. Όσον αφορά τους οργανισμού, οι οργανισμοί που εντάσσονται στην εντολή της DG Sante, είναι η η Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων και η CDC που συνεργαζόμαστε πολύ καλά, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι το δυνατόν καλύτερο. Έχουμε εξάλλου ε, εξασφάλιση για την εφαρμογή των ετησίων, την εκτέλεση μάλλον των ετήσιων λογαριασμών αυτών των τριών οργανισμών. Ε, προσβλέπουμε λοιπόν στην συνέχιση της συνεργασίας μαζί τους και την εξασφάλιση ότι με τους διαθέσιμους πόρους θα καταφέρουμε ό,τι είναι ε, δυνατόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Επόμενα βήματα θα είναι οι τροπολογίες προς κατάθεση μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί και η ψηφοφορία θα γίνει στην Επιτροπή μας στις 21 ε, Ιανουαρίου και στην ΚΟΝΤ στις 9 Φεβρουαρίου. Και από την Ολομέλεια θα περάσει το θέμα τον Μάρτιο. Σας ευχαριστώ όλους τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Αρχίζουμε με το επόμενο θέμα. Εγώ θα χρειαστεί να αποσιάσω. Ζητώ συγγνώμη. Ο Σεπ με αντικαταστήσει στο Προεδρείο και θα δώσω το λόγο στην Κριστιάν Θελτερμόζε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουν μείνει και πολλοί στην αίθουσα, αλλά ε, να σας αναφέρω ότι στην προηγούμενη θητεία προσπαθήσαμε στην Επιτροπή μας να στηρίσουμε μια πρωτοβουλία ΜΚΟ για να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε το ευρωπαϊκό έτος ε, των πρασινότερων, για πρασινότερες μάλλον πόλεις. Αυτό θέλουμε να το ξανασυζητήσουμε πάλι στην Επιτροπή ΕΝΒΗ και η ιδέα είναι να υποστηρίξει η Επιτροπή αυτή την πρωτοβουλία. Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό έτος για πρασινότερες πόλεις, επειδή αυτό έχει να κάνει με τις πρωτοβουλίες μας περί περιβάλλοντος και επειδή αυτό συμβαδίζει και με τις προτεραιότητες. Οι πράσινες πόλεις έχουν μεγάλο ρόλο να παίξουν στην πράσινη μετάβαση. Πρέπει να εστιάσουμε στις πόλεις και στις ε, πράσινες πρωτοβουλίες. Θεωρούμε λοιπόν πως είναι δυνατόν να προωθηθεί η πράσινη μετάβαση, διότι οι πόλεις μας έχουν να παίξουν ε, ρόλο κλειδί. Υπάρχουν πολλοί και διάφοροι λόγοι να εστιάσουμε στις πόλεις και πώς αυτές μπορούν να συμβάλλουν στην πράσινη ατζέντα. Γι' αυτό και προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Έτος για Πρασινότερες Πόλεις. Στο ψήφισμα προτείνουμε το έτος αυτό να είναι το 2021 ε, μπορεί να υπάρξει, ε, υπάρχει μάλλον μια τροπολογία ώστε να αυτό να καθυστερηθεί για το 2022 στο σχεδιασμό για πρασινότερες πόλεις να είναι δυνατός και να μπορέσουμε να εστιάσουμε σωστά στις πράσινες πόλεις. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θέλουμε να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να έχουμε περισσότερους πράσινους χώρους, να εστιάσουμε στην έρευνα μέσα στο πλαίσιο της καινοτομίας να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να κάνουν περισσότερα ώστε η γειτονία να είναι ε, πιο πράσινη και να εστιάσουμε γενικότερα στην πράσινη νοοτροπία ώστε να προωθήσουμε τους, τις πράσινες περιοχές. Υπάρχουν ένα σωρό θετικά στοιχεία σε αυτό το ψήφισμα. Ως συνυπεύθυνη και συνσυντάκτρια αυτού του ψηφίσματος θέλω να ενθαρρύνω την Επιτροπή Περιβάλλοντος να εγκρίνουμε ένα ευρωπαϊκό έτος για πρασινότερες πόλεις για το 2022, γιατί αυτό θα συμβάλλει στην, ε, στο πρασίνισμα των πόλων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ βγαίνω από το ρόλο μου ως γραμματέας, αλλά θα δώσω το λόγο στην κυρία Βλερουά. Ευχαριστώ. <laughs> Mais c'est une confusion tellement fréquente, Madame l'Interprète. Κοιτάξτε, ε, το όνομά μου το είπατε κάπως λάθος, αλλά δεν πειράζει, συχνά μου το μπερδεύουν και καταλαβαίνω τι εννοείται εμένα. Να επιμείνω για το γεγονός ότι οι μεγάλες πόλεις και οι μητροπόλεις είναι σημαντική περιφερειακή ε, ε ε, μοχλή διάδοση των ευρωπαϊκών πολιτικών και τα προβλήματα που σχετίζονται με τα αστική ρήπανση ε, είναι πολύ ε, μεγάλα, γι' αυτό είναι απαραίτητο να επιμείνουμε έτσι ώστε οι πολιτικές του Πράσινου Συμφώνου να διαδίδονται μέσα από τις μεγάλες πόλεις και μητροπόλεις. Merci. Désolé, je continue sur un mode un peu spécial, Σας ευχαριστώ λοιπόν, αλλά πρέπει να συνεχίσω εγώ. Θα μιλήσω στα γερμανικά. Θα ήθελα να σας πω ότι σκέφτηκα όταν ασχολήθηκα με αυτή την έννοια. Εγώ προέρχομαι από μια πόλη που καταστράφηκε κατά 70% στο Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο και που τη δεκαετία του 50 μόνη της ε, ανοικοδομήθηκε. Δηλαδή η εμπειρία μου είναι μια εμπειρία γκρίζας πόλης μάλλον. και εγώ χάρηκα πολύ όταν πήγα στο εξωτερικό και είδα συγκριτικά πράσινες πόλεις. Πέρυσι ασχοληθήκα πολύ με το ζήτημα της βιοποικιλότητας. Φαίνεται ότι πεθαίνουν ε, έντομα σε όλο τον κόσμο και στην Γερμανία. Έχουμε μια καταπληκτική ιδέα ε, συνεργασία ε, δήμων για μεγαλύτερη βιοπικιλότητα. Εκεί έμαθα ότι οι ιδιωτικοί μας κήποι στη Γερμανία στο εμβαδό τους έχουν μεγαλύτερο εμβαδόν από ότι όλοι οι χώροι προστασίας, όλοι οι χώροι φυσικής προστασίας τους Δήμους. Λοιπόν βλέπει κανείς γιατί χρειάζεται μια στρατηγική βιοπικιλότητας και στις πόλεις. Η πόλη είναι το κομμάτι όπου χρησιμοποιούνται λιγότερα να από οπουδήποτε αλλού. Και οι περιοχές αυτές ε, προσφέρονται πολύ καλά για να δημιουργηθούν βιότοποι. Σε πολλές πόλεις, ε, στην ε, Ρινανία, Παλατινάτο υπάρχουν ε, εποχές που υπήρχαν ανέκαθεν μικρά χώροι που θα μπορούσαν να αποτελέσουν ε, hot spot βιοποικιλότητας ε, με τη σωστή ανοικοδόμηση. Και αυτό μα μας ενθουσιάζει τους πράσινους γιατί έχουν και πολύ χαμηλό κόστος και είναι πολύ εύκολο να τα διαχειριστεί κανείς Πρέπει να δούμε επίσης να λάβουμε υπόψη και την ε, ικανότητα αντοχής ε, των πόλεων, των δήμων σε εποχές ε, κλιματικής κρίσης μέσω των ολοένα και, επιδεινούμενων, και περισσότερο επιδεινούμενων καιρικών φαινομένων. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό δίνει μια, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για ένα πανευρωπαϊκό έργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, μια σύντομη παρέμβαση για να πω ότι αυτό το πρασίνισμα των πόλεων είναι κάτι πολύ σωστό. Ξέρετε, με τη μεγάλη μετανάστευση των πληθυσμών το 19ο αιώνα ε, με την, ε, και τη δημιουργία των τεράστιων σιδηρουργικών ε, κέντρων, φτιάξαμε πόλεις ε, που δεν άρμοζαν στον άνθρωπο και η παγκοσμιοποίηση και ειδικότερα η Ευρώπη που θέλησε ένα ειδικό μοντέλο, τις μεγάλες περιφέρειες, τις μεγαλοπόλεις, δεν είναι ουσιαστικά τίποτα άλλο παρά ένα φαινόμενο που ερήμωσε τις ε, εξοχές μας. Φτιάξαμε μεγαλοπόλεις όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο οι ζωές μας να είναι ανθρώπινες. Σε αυτό προσδίθεται το πρόβλημα των υποδομών, οι οικοδομές, ε, η εκένωση των υδάτων, η διαχείριση των υδάτων, των αποχετεύσεων, της ε, κυκλοφορίας. Όλα αυτά γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Το πρασίνισμα των πόλεων, α το πούμε μεταξύ μας φυσικά, δεν είναι παρά το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που θα ήταν καλό θα ήταν να ξαναδώσουμε στις εξοχές μας ε, ε τις ιδιότητες του οικότοπου ε, του καλού μέρους να μένεις που είχαν ανέκαθεν ε, για να μπορέσουμε να, να ε, απαλύνουμε λίγο το, τις δυσκολίες της Μητροπόλης, της Μεγαλοπόλης. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Χόης έχει. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ πολύ. Εγώ δεν έρχομαι από κάποια πόλη που καταστράφηκε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι δικέ μα πόλεις στην Κεντρική Ευρώπη καταστράφηκαν από 40 χρόνια αυταρχικά καθεστώτα αλλά πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό έτος των κέντρων των πόλεων είναι κάτι απαραίτητο για μας, ε, για τις πιο πράσινες πόλεις, για το ευρωπαϊκό έτος των πιο πράσινων πόλεων για να μας βοηθήσει να κάνουμε τις αλλαγές ε, που είναι αναγκαίες ε, για την επιβίωση και για την αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων των κλιματικών και που αφορούν και τη βιοποικιλότητα. Θα μας βοηθήσουν να δείξουμε πώς η πόλη μαζί ελπίζουμε με αυτό το κοινοβούλιο θα ηγηθούν αυτή τη ε, μάχη κατά της ε, κλιματική κρίσης γιατί αυτό ε, από την εμπειρία μου των τελευταίων εβδομάδων παρατηρώ ότι πολλές φορές οι Δήμοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή και υφίστανται τεράστιους μετασχηματισμούς μέρος των οποίων είναι ότι οι υποδομές και οι δημόσιες μεταφορές ε, ότι πολλοί κόσμοι προτιμά πλέον τι δημόσιε μεταφορέ πέρα τι ιδιωτικέ. Ο χώρο ε, στα κτίρια, οι κοινοί χώροι, ε, ο κόσμο ανακτά του κοινού χώρου και του μετατρέπει σε κάτι πιο φιλικό προ τον άνθρωπο. Και ελπίζω φέτο η φετινή χρονιά να αποτελέσει την αφετηρία, όχι μόνο την αφετηρία πολλών πραγμάτων, αλλά να δούμε ήδη πολλά παραδείγματα, πολλά αποτελέσματα που θα εμπνεύσουν και άλλου και στην Ευρώπη και πέραν αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Ριβαζή. Ναι, εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτή την ε, πρωτοβούλια. Πράγματι. Όταν είχαμε ε, το φετινό καλοκαίρι τους καύσονες, οι πόλεις ήταν αυτές που υπέφεραν περισσότερο. Εξού η σημασία του να βάλουμε περισσότερα φυτά στις πόλεις. Για να γίνει αυτό πρέπει να αυξήσουμε και τη βιοπικιλότητα, να φέρουμε δέντρα να βρούμε τρόπους μείωσης της θερμοκρασίας της πόλης. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα δεύτερο ζήτημα, η, η ρήπανση. Και βλέπουμε ότι στις πόλεις η ρήπανση είναι πολύ ψηλή, ειδικότερα όσον αφορά τα μικροσωματίδια. Στη Γαλλία κάτι που έχει προχωρήσει ήταν το εξή. Ε, ένα διάταγμα του 2019 που απαγορεύει τη χρήση ζανιοκτώνων σε πόλεις. Και τώρα έχουμε περισσότερα έντομα στι πόλει, ακόμη και μέλισσε, γιατί κανεί δεν χρησιμοποιεί πλέον ζεζανιοκτώνα. Έχουμε κάτι άλλο που μα ανησυχεί με τη γεωργία, γιατί ξέρετε, ε, θέλαμε εμεί κάποια διατάγματα που να απαγορεύουν ε, κοντά σε ε, σπίτια. Αλλά να σα πω κάτι αντίθετο όμω με αυτή την υπόθεση ε, των περισσότερων φυτών στι πόλει. Η ιστορία του 5G Θέλουμε να φτιάξουμε συνδεδεμένε πόλει και βάσει μια μελέτη που έγινε στην Αγγλία από το Υπουργείο Πολιτισμού και Ψηφιοποίηση, ε, λέγεται ότι αν θέλουμε να εγκαταστήσουμε την τεχνολογία 5G, ε, πολλαπλασιάζουμε, δεκαπλασιάζουμε ουσιαστικά τι κεραίε και θα αντιληφθούμε ότι οι δέσμες ε, της 5G είναι στενές για να μεταφέρουν περισσότερα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι αν βάλουμε φύλλα, δέντρα, μειώνεται η απόδοση κατά 80% ή κατά 70%. Δηλαδή, ε, φύλλα βρεμένα θα μειώνουν την απόδοση του 5G. Δηλαδή, από τη μια θέλουμε να βάλουμε την τεχνολογία 5G, να συνδέσουμε ε, σε μεγαλύτερο βαθμό τι πόλει και από την άλλη θέλουμε να φυτέψουμε δέντρα. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώ θα γίνει όλο αυτό πριν να αρχίσουμε να αναπτύσσουμε την 5G με, σε βαθμό ασταμάτητο ουσιαστικά. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα, η κυρία Βιλάνου Εύα στο Πρόεδρε. Είδαμε χθε ότι άρχισε η COP25 για το κλίμα που είχε προβλεφθεί για τη Χιλή και από τότε που ο πρόεδρος Πινιέρα έκανε πόλεμο στην ε, χώρα του πήγε στην Μαδρίτη η COP24. Βλέπουμε ότι οι πολίτες όλες, είναι, οι είναι αυτοί οι οποίοι καταγγέλουν αυτά τα οποία γίνονται κατά της προστασίας του κλίματος. Βλέπουμε ότι οι ΙΠΑ έχουν φύγει από αυτήν την οργανώση. Θα ξέρουμε ότι παντού θα πρέπει να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του, διοξιδίου του άνθρακος και όπως λέει και Διεθνής Οργανικός Οργανισμός Υγείας πάρα πολλά άτομα πεθαίνουν εξαιτία αυτής της δηλητηρίασης. Πιστεύω λοιπόν ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να κάνουμε κάτι όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, αλλά θα πρέπει να είμαστε ε, να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι 10 πολύ μεγάλες πολυεθνικές στον κόσμο ρηπαίνουν κατά 70% και στην Ισπανία οι εταιρείε μας ένα μεγάλο ποσοστό επιπή. και αυτές είναι αυτές οι οποίες είναι οι χορηγοί της ε, συνεδρίασης της ΚΟΠ αυτή της μεγάλης. Θα πρέπει λοιπόν να μην χρησιμοποιούμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Δεν θα πρέπει να ε, σταματήσουμε εδώ και βεβαίως θα πρέπει ο καθένας προσωπικά να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Τι έχουν να κάνουν οι πολίτες. Όλο και περισσότερο παίρνουν το αυτοκίνητά τους, κάνουν περισσότερα χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάνε στη δουλειά τους. Γιατί, Γιατί και τα νίκια στα κέντρα των πόλεων έχουν αυξηθεί και χρειάζεται να πάνε να μείνουν στα προάστια τα μακριά μακριά από το κέντρο και να γυρίσουν πίσω. Τι γίνεται με το σημερινό μας σύστημα. Επίσης, μικρές ε, ε, εταιρείε και βιομηχανίες κλείνουν και τα γιαούρτια ακόμη που είναι ένα φρέσκο υποτίθεται προϊόν κάνουν πολλές φορές 5 και 10.000 χιλιόμετρα με αυτά στο ψυγείο μας. Θα ήθελα λοιπόν να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι να έχουμε χώρους πρασίνου σε όλες τις πόλεις παντού. Μην ξεχνάμε ότι θα πρέπει να αναγνωρίσουμε όλοι ότι με τον ίδιο τρόπο αναπνέουμε, όπως και να πιστεύουμε ότι κάποια πράγματα είναι σημαντικά στη ζωή. Ευχαριστώ, πιστεύω ότι δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι, γι' αυτό θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιό, από την κυρία Κλάουντια Φούσκο, να μας πει ποια είναι η δική της άποψη για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ που μου δίδει το λόγο και για την πρόταση που κάνετε. Την χαιρετίζουμε. Όντως, πιστεύουμε ότι στο παρόν πολιτικό πλαίσιο οι πόλεις πρέπει επίσης και όλοι οι πολίτες να παίξουν ρόλο σημαντικό για την ε, διόρθωση των ε, κλιματικών προβλημάτων. Το είπε και η κυρία Μόζη. Οι πόλεις είναι επίσης το μέρος όπου όλα τα επίγοντα περιστατικά λαμβάνουν χώρα. Το είπε κάποιος συναδελφός σας. Και αυτό που λένε και πολλοί δήμαρχοι είναι ότι θα πρέπει να μπορούν στι επίγους καταστάσεις να έχουν τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται. Και ανταποκρίνονται. Συμβαίνουν ε, λοιπόν κάποια πράγματα και θα ήθελα να συγχαρώ και κάποιους δημάρχους πόλεων για τον εξαιρετικό ρόλο που διαδραματίζουν στην αντιμετώπιση τέτοιων κατασκοφών. Ξέρουμε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απονέμουμε και ένα βραβείο στην πραγματική πολιτική που έχει σημασία με το έργο που επιτελούν ενεργά κάποιοι δήμαρχοι. Ελπίζουμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε και όλες οι πόλεις θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το Green Deal. Τώρα η βιοπικιλότητα, το πρασίνισμα το πόλεων είναι ακόμη πιο σημαντικό. Θα κάνουμε ακόμη και κάτι παραπάνω. Πιστεύουμε ότι μεταξύ των πρωτοβουλειών προτείνεται να υπάρξει μια κοινοτική στρατηγική βιοπικιλότητας. Και αυτό θα είπαμε ότι θα γίνει στις 100 πρώτες μέρες της ε, ανάληψη της νέας επιτροπής. Και προσπαθούμε να ασχοληθούμε με την βιοπικιλότητα, δεδομένου ότι μας προστατεύει. Επίσης, στα πλαίσια της κινητικότητας πρέπει να μειώσουμε την ε, εκπομπή καυσαερίων και όχι μόνο του διοξείδου του άνθρακος και την ηχορύπανση θα πρέπει να μειώσουμε. Σε μία έκθεση σχετική είδαμε ότι υπάρχουν για, τους πολίτες πολλά δευτερεύοντα καταστροφικά αποτελέσματα. Επίσης χαιρετίζουμε την ιδέα αυτή να αφιερώσουμε ένα έτος στις ε, πιο πράσινες πόλεις. Θα πρέπει βεβαίως να ληφθεί η αποφασία από το σύλλογο των επιτρόπων, διότι θα πρέπει για να είναι επιτυχής αυτή η χρονιά να προετοιμαστεί σωστά. Στην αρχή της παρέμβασης υπενθυμίστηκε ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία ΜΚΟ. Αλλά θα πρέπει να πω ότι και εμείς και να υπενθυμίσω ότι και εμείς ε, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες όχι μόνο με για συνεργασία με τις ΜΚΟ, αλλά όλους τους εμπρεκόμενους φορείς. Γι' αυτό θα θέλαμε να εργαστούμε και πιο ε, στενά και να δημιουργήσουμε και στενότερους δεσμούς με το δίκτυο των, ε, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλουμε να έχουμε χρόνο να επεξεργαστούμε αυτή την τροπολογία. Είμαστε στη διάθεσή σας ούτως ή άλλως για οποιοδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών 10 Δεκεμβρίου 11 το πρωί. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας 20-21 Ιανουαρίου στην Ολομέλεια ψηφοφορία θα λάβει λόγο τον Φεβρουάριο. Ευχαριστώ πολύ. Και περνούμε τώρα στο επόμενο θέμα που είναι ε, τροποποιητική απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον ε, Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το θέμα πριν το παρουσιάσει ο εισηγητής μας, για το θέμα αυτό θα μας μιλήσει ο κύριος, ο, εκ, εκπρόσωπος της Έχει 10 λεπτά. Και μετά θα ακούσουμε τον εισηγητή μας. Πρώτα όμως τον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να παρουσιάσω αυτή την πρόταση σήμερα. Ποια είναι η συλλογιστική. Μάλλον τεχνική και θα ήθελα να μην μπω σε λεπτομέρειες. Γιατί υπευλήθη αυτή η πρόταση. Ένας από τους λόγους είναι τα κονδύλια του PDP και θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί στον ε, φετινό ε, προϋπολογισμό το θέμα αυτό. Στα πλαίσια του PDP τα θέματα αυτά αναφέρονται μαζί με τα θέματα της ασφάλειας. 1,4 δις έχουν δοθεί. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι θα μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τον ε, εξορθολογισμό που έγινε στα πλαίσια του πλαισίου δημοσιονομικού πλαισίου. Έτσι λοιπόν τα πράγματα για ένα τόσο πολύπλοκο ε, θέμα είναι πιο απλά. Κάτι άλλο το οποίο θα ήθελα να αναφέρω, το οποίο είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε, είναι ότι η πολιτική προστασία είναι μία δραστηριότητα από την οποία σχεδόν 100% εξαρτώμεθα από τα κράτη-μέλη μία μη οικονομική πρόταση είναι να μπορέσουν να διαγραφεί το πρώτο προσάρτημα της παρούσας απόφασης, διότι με την αναθεώρηση του συστήματος που θα δημιουργήσει περισσότερα κονδύλια ε, στα κράτη-μέλη και το περίφημο Rescue, ε, αλλάζουν τα πράγματα. Βεβαίως, το θέμα της ετοιμότητας ε, είναι πολύ σημαντικό, γι' αυτό τα ποσοστά πρέπει να παραμείνουν. Επίσης, θα πρέπει να πω ότι αφορούσαν, δεν αφορούσαν πληρωμές, αλλά What counts for υποχρεώσεως καταρχάς. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα. So timetable is therefore uh, that we hope... Έχετε λοιπόν εδώ το χρονοδιάγραμμα. Προσπαθούμε στις αρχές του 2020 να κάνουμε τριμερή διάλογο και δεδομένου ότι δεν προτείνουμε εμείς πλήρως τον προϋπολογισμό για όλες αυτές τις δράσεις θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις μεταξύ των τριών οργάνων σίγουρα για να προχωρήσουμε. Τα πιο σημαντικά σημεία είναι τα εξής. Θα χρειαστούμε την ε, μεγάλη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να μπορέσουμε να έχουμε τον προπολογισμό που θα μας επιτρέψει ε, να συγχρηματοδοτήσουμε τα κράτη-μέλη. Πρώτα απ' όλα ε, για τα ειδικά αεροσκάφη τα τύπου Καναντέρ για τις ε, πυρκαγιές. Επίσης την ιατρική από αέρο νοση ε, δυνατότητα για ασθενείς με πολύ σοβαρές ασθένειες και μολυσματικές όπως ασθενείς που πάσχουν από, έχουν έμπολα. Δεύτερο, Η εκτέλεση του προπολογισμού είναι υποχρέωση για την Επιτροπή και στην πράξη στο σύστημα αυτό έχουμε να κάνουμε με την θέληση των κρατών μελών να δημιουργήσουν πιστώσεις ώστε να αναλάβουμε ε, δραστηριότητες πρόληψης και ετοιμότητας. Χρειαζόμαστε λοιπόν στον σχεδιασμό τον οικονομικό ευελιξία. Μόνον έτσι θα είμαστε σίγουροι ότι όντως μπορούμε να εκτελέσουμε τον προϋπολογισμό σε ποσοστό 100%. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η διαγραφή του προσαρτήματος 1 δεν μειώνει το ποσό το οποίο θέλουμε να δαπανίσουμε για πρόληψη. Προβλέπεται για τον PDP για τέτοιου είδους δραστηριότητες που θεωρούμε ότι είναι το πιο σημαντικό αύξηση ε, κατά 40% των κονδυλίων που έχουν δοθεί στα πλαίσια του ε, παρόντος, όχι του καινούριου PDP. Όλα αυτά τα θέματα συζητούνται και στο Συμβούλιο λεπτομερώς και θα ήθελα πάρα πολύ ε, σύντομα να σχολιάσω τι είπαν. Πρώτα απ' όλα υπάρχει η δυνατότητα να μπορέσουμε διάφορα πολυετή προγράμματα εργασίες να τα παρατείνουμε ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται τώρα δεν επιτρέπει να δαπανηθούν όλα τα κονδύλια ε, για την πρόληψη. Γι' αυτό προβλέπεται η παράτασή τους, για να μην έχουμε αδιάθετα κονδύλια. Αυτό λοιπόν το ζητά το, Συμβούλιο και προτείνουμε εμείς κάτι τέτοιο να υποστηριχθεί ώστε να υπάρχουν πενταετή πίνα. Ε, πολυετή προγράμματα εργασίας, πράγμα το οποίο θα κάνει πιο εύκολες τις δραστηριότητες πρόσληψης. Και... Τώρα, η ευελιξία βρίσκεται εδώ με τα πολυετή προγράμματα εργασίας και με κάτι άλλο που θα επιτρέπει την ε, έμεση διαχείριση. Για ποιο λόγο, διότι θα έχουμε σημαντικότερα, πολύ σημαντικά κονδύλια με πιο πολύπλοκα συστήματα διαχείρισης. Το κράτη-μέλη ε, ζητούν κάτι τέτοιο, κάνουν μειοδοτικούς ε, διαγωνισμούς, γι' αυτό για κάποια κονδύλια πρέπει να επιτρέψουμε αυτό το indirect management. Και επίσης θα πρέπει να επιτρέψουμε να υπάρχει συνεργασία με ερευνητικά κέντρα και με κέντρα αριστείας. Προτιμούν για αυτή την περίπτωση τα κράτη-μέλη να ιδρυθεί μία δωδεκαμελής γραμματεία εδώ. Αλλά ε, εάν ε, συνεχίσουν να ζητούν κάτι τέτοιο για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε στα κράτη-μέλη αυτό το οποίο ζητούν, θα χρειαστούμε περισσότερα κονδύλια. Εδώ βλέπετε κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Κάποιες χώρες όταν ε, το 13, συζητήθηκε η απόφαση 13-13 είναι όταν έχουμε επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Δεξαμενής Πολιτικής Προστασίας, να υπάρχει ε, κάλυψη κοινοτική κατά 25% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν παρενέβησαν οι δικές μας δυνάμεις μετά ε, από την, ε, τον τυφώνα Ίζα στη Μοζαμβίκη δεν είδαμε ότι δεν ήταν η καλύτερη λύση. Είπαμε λοιπόν στην Επιτροπή ότι θα πρέπει για τέτοιου είδους επιχειρήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε πιο γενναιόδεροι δεδομένου ότι η πολιτική προστασία είναι σχετικά φτηνός τρόπος επέμβασης. Είπαμε λοιπόν ότι θα πρέπει να ξεπεράσουμε αυτό το ποσοστό. Και τελικά, μια πιο τελευταία εξέλιξη, την οποία όταν αρχίσαμε να διαπραγματευόμαστε δεν γνωρίζαμε σε όλες τις λεπτομέρειές της, αλλά τώρα την ξέρουμε καλύτερα. Το σύστημα Γαλιλαίο θα χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιηθεί στο μέλλον σε περίπτωση καταστροφής να ειδοποιεί τους πολίτες ή για μια καταστροφή που επίκειται ή για μια που έχει ήδη πέσει στο κεφάλι των πολιτών. Και βεβαίως στα κράτη-μέλη θέλουμε να έχουμε και έναν συντονιστή. Η τροπολογία λοιπόν, η αλλαγή αυτή αφορά ότι οι εθνικές αρχές πολιτικής προστασίας θα πρέπει να μας λένε ποιο είναι το συντονιστικό σημείο, πού θα εστιαστεί αυτός ο συντονισμός, ώστε να έχουμε ένα ιδεατό σύστημα. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ανακράτο μέλος μία διεπαφή ε, επιχειρησιακή για να βοηθούμεθα σε περίπτωση, για να συνεντώνει μέσω Γαλιλαίο, για να βοηθούμεθα σε περίπτωση καταστροφών. Συμπερασματικά, θα κάνω στην Επιτροπή σας έκκληση να κατανοήσει ότι φέτος δώσαμε, έχουμε επιστρέψει 45 εκατομμύρια ευρώ διότι δεν μπόρεσαν τα κράτη-μέλη έγκαιρα να ε, χρησιμοποιήσουν τις πιστώσεις. Θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη και θα τους δώσουμε αρχές του επόμενου έτους προθεσμίες για να μας πούνε ποιος είναι ο σχεδιασμός τους για τα επόμενα χρόνια, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε εκτέλεση του προϋπολογισμού σε ποσοστό 100%. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να το κατορθώσουμε αυτό και φέτος επειδή είχαμε λιγότερους μήνες, το ότι δεν μπόρεσαν να εκτελεστούν όλα τα κονδύλια που προβλεπόνταν, δεν θα θεωρηθεί ως κάτι το οποίο πρέπει να επαναλάβουμε τα επόμενα χρόνια. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ λογικοί. Είδατε φέτος το καλοκαίρι τι έγινε και εντός Ευρώπης και εκτός. Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε κάθε ευρώ μέσα από αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό πρέπει να ενεργούμε και έγκαιρα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Ε, ναι. Είπατε ότι είναι επιφανειακό, αλλά ε, μπορεί έτσι να έχουμε μια καλή εικόνα περί τίνος πρόκειται. Και όπως σας είπα, είναι ένα από αυτά τα θέματα στην προστασία, ε, την πολιτική που δεν συζητάμε αρκετά συχνά. Είναι όμως ένα πολύ σημαντικό έργο που κάνει η δική σας μονάδα και που εμείς πρέπει να εποπτεύουμε. Μα δώσατε μια πολύ καλή εικόνα. Σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Ανδρουλάκη, ώστε να μας δώσει τη δική του γνώμη και την αρχική του απάντηση σε σχέση με αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θέλω να επαναλάβω τα όσα ήδη αναφέρθησαν ε, από την Επιτροπή στην παρουσίασή της. Ε, συμμετείχα και στις προηγούμενες διαπραγματεύσεις ως ε, σκιώδης ε, εισηγητής. Ε, σίγουρα ήταν δύσκολες διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Καταφέραμε όμως να διασφαλίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τα απαραίτητα εργαλεία για να αντιμετωπίσει τις ολοένα και αυξανόμενες φυσικές καταστροφές αλλά και κάθε νέο είδους απειλές ε, που εμφανίζονται. Συγκεκριμένα, παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που είχαμε με το Συμβούλιο, καταφέραμε να δημιουργήσουμε το RescueU, μια ευρωπαϊκή δεξαμενή μέσων που θα αγοραστούν μεν από τα κράτη-μέλη, αλλά με πολύ μικρό ποσοστό, μάλλον με πολύ μεγάλο ποσοστό συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που κυμαίνεται από 80 έως 90% και θα μπορεί να φτάσει ακόμη και 100% για συγκεκριμένες δυνατότητες. Τα μέσα αυτά θα ανήκουν στα κράτη-μέλη, αλλά η αποστολή τους δεν είναι μόνο εθνική υπόθεση. Αν κριθεί ότι ένα κράτος μέλος χρειάζεται βοήθεια, τότε θα είναι πάντα έτοιμα να ανταποκριθούν. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούμε ένα νέο επίπεδο προστασίας ευρωπαϊκά, διασφαλίζοντας ότι καμία χώρα δεν θα μείνει αβοήθητη. Επιπλέον, δώσαμε για πρώτη φορά τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την επισκευή των εθνικών μέσων που διαθέτουν, εντάσσοντάς τα και αυτά στην εθελοντική δεξαμενή. Δυστυχώς, δεν μπορέσαμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις αρμοδιότητες που θα θέλαμε στο επίπεδο της πρόληψης και του ελέγχου των σχεδίων προστασίας από φυσικούς και άλλους κινδύνους. Παρόλα αυτά, συμπεριλάβαμε μια δικλίδα ασφαλείας, ώστε σε περίπτωση συχνής ενεργοποίησης του μηχανισμού από κάποιο κράτος μέλος, η Επιτροπή να μπορεί να εξετάσει τα μέτρα πρόληψής του και αν χρειάζεται να προβαίνει σε συστάσεις για τη λήψη επιπλέον μέτρων από το κράτος αυτό. Από το Μάρτιο, οπότε και μπήκε σε εφαρμογή το νέο αυτό πλαίσιο, έχουμε δει ήδη τα πρώτα θετικά αποτελέσματα. Έξι χώρε συμμετέχουν στην προσωρινή δεξαμενή γιού, που δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό μέχρι να αγοραστούν οι νέες δυνατότητες. Είδαμε μάλιστα την πρώτη ενεργοποίησή του κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού από τη χώρα μου, τη χώρα που προέρχομαι την Ελλάδα, για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που ξέσπασαν στην Εύβοια κατά τον Αύγουστο. Επίσης, η λίστα με τα μέσα που θα πρέπει να αγοραστούν για τον εξοπλισμό του Rescue δεν περιορίζεται μόνο στα ενέργεια μέσα δασοπυρόσβεσης, αλλά έχει και ιατρικές μονάδες για την αντιμετώπιση έκτακτων ιατρικών περιστατικών και επιδημιών. Με αυτή την πρότασή μας και που παρουσίασε πριν από λίγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή που μας παρουσίασε, στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το εργαλείο αυτό αλληλεγγύης που δημιουργήσαμε θα έχει όλα τα απαραίτητα μέσα για να λειτουργήσει. Η πρόταση της Επιτροπής για ένα προϋπολογισμό 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ την περιοδο 2021 2021-2027 μας βρίσκει απολύτως σύμφωνος και θα την υπερασπιστούμε στις διαπραγματεύσεις που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Είναι μια επένδυση για το μέλλον, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και την όξυση των καιρικών φαινομένων, προστατεύοντα αποτελεσματικά του πολίτε τη. Είναι επιπλέον μια καλή ευκαιρία να διορθώσουμε δυσλειτουργίε που παρουσιάστηκαν, καθώς και κάποια ζητήματα που δεν είχαμε λύσει την προηγούμενη, κατά την προηγούμενη αναθεώρηση. Έχοντας δει τη μερική γενική προσέγγιση του Συμβουλίου, έχω να παρατηρήσω ότι είναι θετική η πρόβλεψη για κάλυψη των εξόδων των μέσων που ανήκουν στην εθελοντική δεξαμενή, αλλά δραστηριοποιούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να είμαστε σε θέση να προσφέρουμε τη συνδρομή μας τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ επίσης πολύ θετική τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το δορυφορικό σύστημα Γαλιλαίος για την αποστολή μηνυμάτων εκτάκτης ανάγκης στους πολίτες που βρίσκονται σε κίνδυνο. Πιστεύω βέβαια ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο στην παροχή της δυνατότητας, αλλά οφείλουμε να αναγκάσουμε, τουλάχιστον να πιέσουμε, το σύστημα αυτό να αξιοποιηθεί από όλα τα κράτη-μέλη. Και το λέω αυτό διότι έχω το παράδειγμα το αρνητικό της χώρας μου, που είναι μια άσχημη εμπειρία για το συγκεκριμένο θέμα, όπου μετά από πολλά χρόνια και διάφορες εξαγγελίες ότι το σύστημα αυτό παραμένει ε, θα ενεργοποιηθεί, το σύστημα αυτό παραμένει ανενεργό και δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν οι πολίτες ενώ έχουμε πολλές φυσικές καταστροφές. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε και στη συνέχεια όταν παρουσιάσω και το σχέδιο έκθεσης στις αρχές τη επόμενη χρονιά. Είμαι σίγουρος ότι με τη συνεργασία των συναδέλφων από τις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες θα διαμορφώσουμε ένα κείμενο που θα διασφαλίζει ότι ο νέο μηχανισμός πολιτικής προστασία θα είναι αποτελεσματικό, θα έχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες να είναι ασφαλείς σε όποιο κράτος μέλος και αν κατοικούν. Ευχαριστώ. Um, I believe we don't... Πιστεύω ότι δεν έχουμε εκπρόσωπο νούνο μέλο λείπει από το ΕΛΚ. Δεν ξέρω αν κάποιος άλλος από το ΕΛΚ θα πάρει το λόγο εκ μέρους του. Όχι. Ε, ε, για να κάνουμε ένα γύρο των ομάδων. Στέβεν Ιούτε από το Ρινιού. Χαίρετε. Εγώ εδώ είμαι σκιώδης ε, εξ του Ρινιού. δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για αυτό το θέμα. Πότε πρέπει να εγκρίνουμε, να λάβουμε απόφαση και έπειτα συμφωνώ ότι για την υπόλοιπη Ένωση και για τον μηχανισμό προστασίας θα πρέπει να γίνει σημαντική συζήτηση στο πλαίσιο του PDP, διότι έχω την αίσθηση ότι αυτό που έχουμε εδώ είναι ψίχουλα είναι πολύ λίγα, ενώ οι κρίσεις ε, ε, είναι αλλεπάλληλες και μάλιστα επανέρχονται δρυμύτερες και κάθε φορά πρέπει να ψάξουμε δύο ελικόπτερα δεξιά, τρεις ε, ταξιαρχίες θελοντών αριστερά και πάει λέγοντας οι κρίσεις, οι πήγουσε καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις ανακύπτουν διαρκώς και οι Ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν κάτι πολύ πιο συνεπές με ισχυρό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εγώ θα ενημερώσω τα μέλη για το χρονοδιάγραμμα, γιατί ξέρω ότι ε, ε, δεν είναι εδώ οι θα έχουν την δυνατότητα και, και, η Κομισιόν βέβαια θα σχολιάσει μετά. Να σας πω ότι 10 Δεκεμβρίου στις 11 ε, το πρωί είναι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Α, όχι, όχι, λάθος, λάθος, τελείωσα, στάπα. Δύο λεφτά. Κοίταζα... Ε, το χαρτάκι του Προέδρου από το προηγούμενο θέμα. Λοιπόν, αγνοήστε το. Πάντω, 10 Δεκεμβρίου είναι ημερομηνία, αλλά είναι η ημερομηνία για το σχέδιο έκθεση. Το σχέδιο έκθεση είναι έτοιμο στι 10 Δεκεμβρίου. Μετά θα εξετάσουμε το θέμα στι 20 και 21. 20-21 Ιανουαρίου 2020. Λοιπόν, μην δίνετε σημασία. Α, η Μαργαρίτα δεν είναι εδώ, οπότε η Σίλβια Σαρντώνη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Το σύστημα πολιτικής, ευρωπαϊκό σύστημα πολιτικής προστασίας παρουσιάζεται ως ένας τρόπος να δείξουμε αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Όμως εγώ έχω κάποιες ε, επικρίσεις. για να καταλάβω λοιπόν το εξής. Εγώ εγώ το κράτος δίνω χρήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αγοράσει ελικόπτερα και να προσφέρει κατάρτιση που ίσως μετά να συγχρηματοδοτήσει τη δική μου, ε, τη δική μου χώρα. Ε, εγώ για την Ιταλία έχουμε ήδη πολιτική προστασία και μάλιστα ε, είμαστε σε επίπεδα αριστείας, δηλαδή πληρώσουμε πολύ περισσότερα μου φαίνεται από ότι αν το αγοράζαμε μόνο μας το ελικόπτερο. Τώρα αν θέλει να κάνει πείραμα η Ευρώπη, άλλη υπόθεση. Τώρα και κάτι ακόμα για τις αρμοδιότητες που δεν κατάλαβα. Εγώ λοιπόν από όσο γνωρίζω η αρμοδιότητα για την πολιτική προστασία παραμένει στα κράτη. Για να καταλάβω λοιπόν καλύτερα, αν εγώ η, Ιταλία χρειάζομαι, πρέπει να ζητήσω σε εσά τα μέσα. Μου φαίνεται πως αυτό είναι τρελό. Και έπειτα, Εάν υπάρχουν διάφορα κράτη που κινδυνεύουν, ποιο έχει την προτεραιότητα και ποιο επιλέγει σε ποιον θα δώσει προτεραιότητα για τι ε, παρεμβάσει. Γιατί αν κρίνουμε από το πώ προχωράει η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου θα πρέπει πάντοτε εγώ στην Ιταλία να ελπίζω ότι δεν θα προηγηθεί μια κλιματική κρίση στη Γαλλία και στη Γερμανία πρώτα. Γιατί σίγουρα εγώ ως Ιταλία θα έρθω μετά. Θα ήθελα να ξέρω λοιπόν πώς θα λειτουργήσει ένα τέτοιο σύστημα και από οικονομική άποψη και από άποψη εθνικής ιεραρχίας. Νομίζω πως ε, η δική μου χώρα θα βγει πολύ χαμένη. Ευχαριστώ. Ο Αλεξάνδρ Φόντουλ δεν τον βλέπω. Οπότε θα προχωρήσω στην κυρία Κονέτσνα από την ΚΟΕ. Α, ούτε και εκείνη. Α, είστε εδώ. Είστε εδώ, αλλά δεν θέλετε το λόγο. Εντάξει. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Ναι, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ είμαι μέρος ε, της ε, πολιτικής προστασίας της περιοχής ε, από την οποία προέρχομαι. Λέω κύριος Ντρεώστο και άρα μιλώ εν γνώση των πραγμάτων. Θέλω να σας πω το ποια είναι η λογική μου. Η Ιταλική πολιτική προστασία δημιουργήθηκε το 1976 μετά από τον σεισμό που χτύπησε το Φριούλι Βενέτσια Τζούλια την βορειοδυτική περιοχή. Ο τότε ο αρμόδιος υπουργός Τζαμπερλέτη διάρθρωσε αυτό το κίνημα το οποίο οποίο προήλθε αυθόρμητα από τους πολίτες και από τις ΜΚΟ μέσα από ένα συντονισμένο σύστημα το οποίο μετά μετατράπηκε σε εθνική πολιτική προστασία όπως, όπως έλεγε σωστά η συνάδελφος Σαλντόνε αναγνωρίζεται στην αριστεία του διεθνώς. Δεν περιμένουμε δηλαδή να μας καλέσουν από κάπου για να πάμε. Η προστασία, η πολιτική προστασία η Ιταλική όταν γίνει σεισμός, όταν γίνει οποιοδήποτε θεομηνία και την προ... προάλλες πήγαμε στην Αλβανία, πριν από λίγο είχαμε πάει στην Ελλάδα. Ε, και κάθε φορά ξεκινάμε από μόνοι μας, είμαστε αυτόνομοι. Είναι λοιπόν μια αριστεία που θα έλεγα ότι ευνοείται ή όχι από το γεγονός ότι η σεισμική και η γεωλογική κατάσταση της χώρας μας μας οδηγεί στο να βελτιωνόμαστε χρόνο με το χρόνο και γι' αυτό και πήρα το λόγο. Αυτό έκανε και η συνάδελφος Αλντών εξάλλου. Δηλαδή από τη μια άποψη μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει συντονισμός σε υπερεθνικό επίπεδο γιατί όχι, όμως ανησυχία μας είναι ότι θα αρθεί η λειτουργική μας αυτονομία, η οποία είναι απολύτως απαραίτητη για να είμαστε αποτελεσματικοί. Σήμερα η εθνική πολιτική προστασία με συγκεκριμένα κέντρα που παρεμβαίνουν, που, μάλλον που δίνουν οδηγίες για παρεμβάσεις σε θεομηνίες και φυσικές καταστροφές, το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα και πολύ ε, λειτουργικά. Δεν θέλουμε λοιπόν αυτό να υποσκαπτεί από κάποια ε, ε, διακρατική απόφαση. Κάτι ακόμα και κλείνω, κάτι που που είναι πολύ σημαντικό γιατί εδώ είμαστε σε ένα πλαίσιο όπου συχνά δεν αναφερόμαστε στο κόστος αλλά μόνο στους θετικούς απολογισμούς. Η εθνική πολιτική προστασία κατά 80% αποτελείται από θελοντές, δηλαδή ανθρώπους που δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ για τα όσα κάνουν. Μπορεί να αφιερώσουν δηλαδή τις διακοπές τους ή από δική τους πρωτοβουλία πάνε και βοηθούν αυτούς που έχουν δυσκολίες. Δηλαδή, οποιαδήποτε ε, πολιτική προστασία ε, διεθνής, κρατική θα πρέπει να γίνει στο ίδιο πλαίσιο. Η αλληλεγγύη που είναι μια λέξη πολύ της μόδας αυτούς τους καιρούς ε, στην, ε, στο Κοινοβούλιο δεν μπορεί παρά να εκφράζεται δωρεάν σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών. Ευχαριστώ. Do you have any... Uh, Κύριε Ανδρουλάκη, εσείς θέλετε να κλείσετε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Καταρχάς, στην Ολομέλεια του Μαρτίου θα υπάρξει ψήφιση και το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων. Αυτό για το χρονοδιάγραμμα. Επίσης θέλω να πω το εξής. Το Rescue δεν θα αντικαταστήσει τα εθνικά μέσα πολιτικής προστασίας, ούτε του μηχανισμού που έχει το κάθε κράτος. Και πρέπει να θυμηθούμε γιατί έγινε το Rescue. Διότι το 2017 η Πορτογαλία ζήτησε βοήθεια από τα κράτη-μέλη και κανείς δεν συνεισέφερε τη βοήθειά του. Και είχαν πυρκαγιές με 100 νεκρούς. Και τότε ο πρόεδρος Γιούνκερ και προς τιμή του είπε ότι δεν μπορούμε να στέλνουμε συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο, ναι, για τη λέξη αλληλεγγύη, που δεν είναι θέμα μόδας ή όχι μόδας, είναι ανθρώπινη ανάγκη η αλληλεγγύη και εντός της Ευρώπης και εκτός της Ευρώπης. Και έτσι λοιπόν διαμορφώσαμε την κοινή δεξαμενή μέσων που φιλοδοξούμε να βρούμε τα χρήματα αυτό το 1,4 δις για να έχει πλήρη δυνατότητα όποιο κράτος μέλος όσο ισχυρό ή ανήσιο κι αν είναι και ζητήσει τη βοήθεια αυτή να μπορούμε να την παρέχουμε. Αυτό θα είναι το ρεσιού και αυτό θα είναι ο στόχος των διαπραγματεύσεων που θα προσπαθήσουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιτύχουμε στο μέγιστο βαθμό. Θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο. Σίγουρα υπάρχουν και προβλήματα. Και τα γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όσοι ασχοληθήκαμε το φάκελο και το προηγούμενο διάστημα. Πολλά από αυτά τα αντιμετωπίσαμε, αλλά όχι. Θέλω να σας φέρω το παράδειγμα του κόστους. Ξέρετε, και το λέω για τους νέους ευρωβουλευτές, ότι υπήρχε μέσα στις διαπραγματεύσεις να πληρώνει και ένα κομμάτι της χρήσης το κράτος μέλος μετά από μία περίοδο περισσότερων χρήσεων από όσες θα μπορούσε να δικαιούται. Νομίζω την τρίτη χρήση. Το απαλείψαμε αυτό, ώστε να μην πληρώνει καθόλου, να μην έχει κόστος. Άρα κάποια θέματα, αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνει σωστές διαπραγματεύσεις, μπορούμε να τα πετύχουμε και αυτός ο μηχανισμός να είναι ένα πραγματικό εργαλείο αλληλεγγύης για τους λαούς της Ευρώπης και ένα μήνυμα ότι όσο πιο πολλά εργαλεία ενοποιητικά έχουμε, τόσο καλύτερη ευημερία θα έχουμε στο μέλλον. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ και τέλος λοιπόν, θα, ζητήσουμε ξανά το, θα δώσουμε ξανά το λόγο στην Κομισιόν αλλά πρώτα ο κύριος Λούχνερ θα μπορούσατε να απαντήσετε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κάτι που ξέχασα Είναι και δράτω τη ευκαιρία που μου δώσετε το λόγο. Σας καλώ όλους ατομικά ή ω ομάδα να έρθετε στο κέντρο συντονισμού απόκρισης έκτακτης ανάγκης. Εδώ δίπλα στη Ρίντα για πιο εκτενή συζήτηση και εξηγήσει. Κάτι που ήθελα να σας εξηγήσω είναι ότι όπως είπα στην αρχή πρόκειται για μεικτή αρμοδιότητα. Συγγνώμη, είναι υποστηρικτική αρμοδιότητα, επικουρική αρμοδιότητα. Ε, δεν τίθεται ζήτημα δημιουργίας κάποιας υπερεθνικής ε, δύναμης. Επίσης, ήθελα να υπογραμμίσω ότι για αυτά που είπαν οι Ιταλοί ε, βουλευτέ. Πράγματι, το, πολιτικό, το σύστημα πολιτική προστασία τη Ιταλία είναι άριστο. Το ίδιο είναι και τη Γαλλία και τη Ισπανία. Ωστόσο, σε κάποιε περιπτώσει, και όχι μόνο πέντε χρόνια, κάθε πέντε χρόνια, πολύ συχνότερα οι χώρε ζητούν αυτέ αμοιβαία συνδρομή, διότι δεν μπορούν μόνε του να αντιμετωπίσουν κάποια καταστροφή. Δείτε μία χώρα, για να σα δώσω ένα παράδειγμα, στι δασικέ πυρκαγιέ που δεν ζήτησε ποτέ ιδιαίτερη αρρωγή ήταν η Κροατία. Αν δείτε το μέγεθο του στόλου τη Κροατία, ό φαίνεται να είναι που φαίνεται να είναι ο στολο το κατάλληλο μέγεθο για να καλύψει οτιδήποτε ουσιαστικά, για να έχει στο ίδιο επίπεδο διασφάλιση στην Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ελλάδα, στην Πορτογαλία, θα έπρεπε να αγοράσει περίπου 65 επιπλέον αεροσκάφη. 40 εκατομμύρια έχουν το ένα. Οπότε ακριβώς είναι, αυτό είναι ακριβώς το θέμα, να εξοικονομήσουν χρήματα όλες οι χώρες δημιουργώντας μια ευρωπαϊκή εφεδρεία που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε από τις χώρες, όχι η ιδιοκτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η ιδιοκτησία των κρατών μελών μας. Έτσι λοιπόν, όταν η Σουηδία χρειάζεται βοήθεια, ε, υπάρχουν πυρκαγιές ε, στο Νότο, ο κίνδυνος ε, ε, αν είναι για παράδειγμα στον Νότο μικρός ο κίνδυνος πάνε τα Ιταλικά αεροσκάφη στη Σουηδία. Άλλε φορέ έχουμε στον Νότο ε, ε, κίνδυνο τόσο υψηλό που καμία χώρα δεν μπορεί να δανείσει αεροσκάφη στην άλλη. Και δεν υπάρχει εφεδρεία. Σε τέτοιε ακραίε καταστάσει πιστεύουμε ότι είναι προτιμότερο να υπάρχουν 10 με 16 αεροσκάφη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συγχρηματοδοτούμενα, να είναι τοποθετημένα κάπου στα κράτη-μέλη και αυτά τα αεροσκάφη θέλω να υπογραμμίσω θα είναι επιπλέον των εθνικών ε, στόλων. Δεν μιλάμε να φτιάξουμε εθνικούς στόλους ε, με ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτή είναι η μία περίπτωση. Μία άλλη περίπτωση είναι το σενάριο όπου τα κράτη-μέλη, ένα κράτος μέλος δεν έχει δικά του μέσα. Κανένα κράτος μέλος στην Ευρώπη. Δεν έχουμε πολιτική αρχή για κινητά νοσοκομεία. Η Ιταλία θέλει να φτιάξει ένα. Εμεί θέλουμε να το υποστηρίξουμε, διότι οι καταστροφέ ευρεία κλίμακα υπάρχει περίπτωση να συμβούν και μπορεί σε τέτοια περίπτωση να χρειαστούμε τέτοιου είδου νοσοκομεία. Κανεί ε, στην Ευρώπη δεν αγοράζει αεροσκάφο με το οποίο μπορεί να εκενώσει ανθρώπου ε, με υψηλά επίπεδα μόλυνση. Γιατί? Διότι η πιθανότητα να συμβεί κάτι τέτοιο, να χρειαστεί εκένωση ανθρώπων με έμπολα ή άλλε τέτοιε ασθένειε, είναι σχετικά μικρή. Αν ωστόσο συμβεί, ο κίνδυνος ε, εκτενούς καταστροφής είναι υψηλότατος αν δεν έχει τα απαραίτητα μέσα. Έτσι λοιπόν η απόφαση να υπάρξει αυτή η αγορά και να γίνει συλλογικά μέχρι το ευρωπαϊκό Προπολογισμού και πάλι όπως είπα με μέσα που είναι ιδιοκτησία των κρατών μελών στη, βασίζεται στην προοπτική που είχαμε εμείς. Τι θα κάνουμε ως Ευρώπη ώστε να είναι φθηνότερο για τα κράτη-μέλη να διαθέτουν ένα αποτελεσματικό σύστημα και όχι για να κάνουμε τα πράγματα πιο ακριβά βάζοντα τον καθένα να αγοράσει τα δικά του μέσα που μπορεί να χρειαστεί και μπορεί να μην χρειαστεί παρά μόνο σε ακραίε περιπτώσει. Οπότε το θέμα είναι, επαναλαμβάνω, επιμερισμό ε, πόρων και ευθυνών. Ε, ευθυνών. Φαίνεται να είναι πολλά χρήματα, αλλά αυξάνει την, ε, είναι επιμερισμό και των χρημάτων και αυξάνει την ασφαλεία των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσουμε. Το σχέδιο εκθέση θα πρέπει να είναι έτοιμο μέχρι τι 10 Δεκεμβρίου. Οι συνάδελφοι τότε θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν το περιεχόμενο σε αυτή την Επιτροπή 20 και 21 Ιανουαρίου. Η προθεσμία και τροπολογίες είναι 28 Ιανουαρίου στις 11 το πρωί και μετά θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή μας στις 5 Μαρτίου και στην Ολομέλεια στις 30 Μαρτίου. Έχετε ερώτηση για διευκρίνηση? Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πολύ σύντομα μια διευκρίνηση και να απαντήσω. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν. Υπήρξε αρκετά κατανοητός. Ε, μας, απάντησε, μας έδωσε απαντήσει σε πολλά κενά που βρίσκουμε στο έγγραφο. Ε, ωστόσο, για τον εισηγητή θέλω να πω Προφανώ δεν έχει ενημερωθεί επαρκώ διότι τον Αύγουστο του 2018 η Ιταλία διέθεσε στην Πορτογαλία δύο Καναντέρ και παρά ε, το γεγονό ότι η Ιταλία παρά το γεγονό ότι η Ιταλία, όπω είπε ο εκπρόσωπο τη Κομισιόν, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα περκαγιών όπω όλε οι χώρε τη Μεσογείου. Οπότε θα ήθελα κάποια διευκρίνηση γι' αυτό, γιατί μιλάμε για ένα επιχείρημα ιδιαίτερα σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μην υποτιμάμε και την δέσμευση των διαφορών χωρών σε αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε. Μια... Yeah, Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Προφανώ έχουμε... έχει γίνει τώρα η συζήτηση, εντάξει, τώρα είναι μια ευκαιρία να, να συμβάλλει ο καθένα να συνεισφέρει κάπω ο εισηγητή. Θέλει πολύ σύντομα τον τελευταίο λόγο για να λυθεί η παρανόηση, αλλά θα έχουμε ευκαιρίε ε, να συζητήσουμε και να αλλάξουμε το περιεχόμενο του κειμένου ε, αργότερα. Παρακαλώ. Πείστε το κουμπί για το μικρόφωνο. Είπα για την καταστροφή το 2017 όταν πέθαναν 100 άνθρωποι, όχι το 2018. Ευχαριστούμε πολύ. Μας βεθάτε Ήταν καλή διευκρίνηση. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, να πω στους συναδέλφους ε, ότι έχουμε εδώ να καλωσορίσουμε κάποιους ανθρώπους. Έχουμε μια, κάποιους επισκέπτες από μέλη τοπικών κυβερνήσεων, ε, επίδοξα μέλη τοπικών κυβερνήσεων από τη Ρουμανία. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστούμε που ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να αντιληφθείτε ότι ε, εργαζόμαστε πολύ συνεργατικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, αλλά οι σχέσει μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι κρίσιμη σημασία. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που είστε εδώ και είστε ευπρόσδεκτοι, πραγματικά. Ένα χειροκρότημα. Πριν προχωρήσουμε. Λοιπόν, τώρα πάμε στο σημείο 31. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με το έγγραφο εργασίας που αφορά την αξιολόγηση ε, της ε, νομοθεσίας της Ένωσης για το αίμα του συστούς και τα κύτταρα. Έχουμε μια παρουσίαση από την Κομισιόν για να ξεκινήσουμε, αν δεν κάνω λάθος, και θα ήθελα να καλέσω τον αναπληρωματικό διευθυντή, Γενικό Διευθυντή της DG Sante, τον κύριο Μαρτινσέσο, να μας παρουσιάσει αυτό το σημείο και για όποιον αναχωρεί παρακαλώ να αποχωρείτε γρήγορα και ήσυχα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Λοιπόν, πριν μπούμε στην αξιολόγηση και στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καλό θα ήταν να, να υπενθυμίσουμε για μια στιγμή τις θεραπείες και του ασθενεί προς του οποίου απευθύνεται και στου οποίου εφαρμόζεται αυτή η νομοθεσία. Η νομοθεσία για το αίμα πρώτα απ' όλα καλύπτει την ασφάλεια και την ποιότητα για αυτή τη στιγμή περίπου 25 ε, εκατομμυρία μεταγγίσεις ε, ερυθρά κύτταρα το χρόνο. Ε, περιλαμβάνουν ερυθρά κύτταρα αλλά και πλάσμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ίδια νομοθεσία καλύπτει την ασφαλή συλλογή 8 εκατομμυρίων λίτρων πλάσματο ετησίω και το πλάσμα είναι σημαντικό υλικό ε, κατασκευής ε, πολύτιμων ιατρικών προϊόντων. Αυτό η νομοθεσία καλύπτει τρεις ε, ομάδες θεραπείων, τρεις τύπους. Πρώτα, τα βλαστοκύτταρα ε, που λαμβάνονται από το μεδουλί και κάθε χρόνο 35.000 ασθενείς στην Ευρώπη χρειάζονται τέτοιες μεταγγίσεις, ειδικότερα ε, για την αντιμετώπιση καρκίνων του αίματος. Η δεύτερη ομάδα για την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή ε, βοηθάμε ομάδες με προβλήματα Έχουμε σχεδόν 800 κύκλους ε, θεραπείας ετησίω, ε, Μιλάμε για αντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων, ε, ας πούμε ανάπλαση δέρματος για ασθενείς που έχουν υποστεί εγκαύματα. Αυτή η νομοθεσία διασφαλίζει την ασφάλεια και την ποιότητα των υλικών για τα ιατρικά προϊόντα. Um, just to recall a bit να υπενθυμίσω λίγο ιστορικά τα κράτη-μέλη έδωσαν εντολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον τομέα μετά από μια τεράστια κρίση υγεία στη δεκαετία του 80 και του 90 που λέω πως σας θα θυμάστε τη μετάδοση του HIV και της υπατήτηδας μέσω μεταγγίσεων και παραγωγών του πλάσματος. Εκείνη την εποχή μεταδόθηκαν και άλλες ασθένειες όπως η κρότης και κύτταροθεραπείες ε, ε, μέσω κυδεροθεραπείων και μεταγγίσεων. Ε, ως απόκριση σε αυτή την κατάσταση τέθηκε σε ισχύ η νομοθεσία. Αλλά όχι μόνο γι' αυτό ε, τελικά θεσπίστηκαν στο άρθρο 168 της Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ αυστηρές ρυθμίσεις για τις διαδικασίες αυτές. Και τα δύο ευρωπαϊκά πλαίσια για το αίμα και για τους ιστούς και τα κύτταρα ε, θέσπισαν ε, υψηλά πρότυπα ασφαλείας ε, και ποιότητας. Τα ηθικά ζητήματα ανήκουν σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας στα κράτη-μέλη. Οπότε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία καλύπτει την ασφαλή και την ποιότητα και αυτά τα πρότυπα καλύπτουν όλα τα βήματα από το σώμα του δωρετή μέχρι το σώμα του παραλήπτη. Μιλάμε για την ε, δωρεά, για τον έλεγχο, τη συλλογή, τη διαδικασία, την επεξεργασία, την αποθήκευση και την αποστολή. Η... Είχαμε τα πρώτα πρότυπα στην οδηγία του 2002 του 1998 και μετά στην 2004 καθώς 23. Κάποιοι από εσάς μπορείτε να είστε δωρητές αίματος και μπορεί να γνωρίσετε τα πρώτα βήματα, αλλά αξίζει να υπενθυμίζουμε τα επακόλουθα βήματα που αποκτούν όλο και μεγαλύτερη σημασία τώρα πηγαίνοντας στην αξιολόγηση αυτή καθ' αυτή, Το βασικό ερώτημα που προσπαθούμε να απαντήσουμε στην αξιολόγηση είναι κατά πόσο αυτές οι οδηγίες που τώρα είναι 15 ετών εξακολουθούν να ε, ε, πληρούν ε, το σκοπό για τον οποίο φτιάχτηκαν. Αν διασφαλίζουν δηλαδή την ασφάλεια και την ποιότητα για τις θεραπείες αυτές. Επίσης εξετάζουμε το κατά, την καταλληλότητα, αλλά πέραν τη καταλληλότητα κατά πόσο θα είναι κατάλληλη και για το μέλλον δεδομένων των τεχνολογικών πρόοδων. Για να απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, συλλέξαμε αποδεικτικά στοιχεία για δύο χρόνια, πραγματοποίησαμε δημόσια διαβούλευση με πάνω από 200 απαντήσεις, με συμμετοχή όλων των μέγιστων των μιζωνών ενδιαφερομένων. Κάναμε πολλές συζητήσεις με ενώσεις ασθενών, δωρητών, ε, επαγγελματικά επιμελητήρια και ενώσεις της βιομηχανίας. Μιλάμε συχνά με τους οργανισμούς, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πρόληψης και Ελέγχου, καθώς και με συναδέλφους από την Κομισιόν και από την USFDA. Έχουμε διαβάσει όλες τις παλιότερες εκθέσεις, ε, καταγγελίες και ερωτήσεις ε, για την Κομισιόν. Έχουμε κάνει και μια εξωτερική μελέτη για επιπλέον πληροφορίε, ε, βιβλιογραφία, συνεντεύξει, έρευνε κτλ. Και επίση έχουμε καλέσει όλου του ενδιαφερομένου για ανταλλαγή απόψεων. Η τελευταία εκδήλωση έλαβε χώρα στι 28 Οκτωβρίου. Και τα... υπήρχε και συμμετοχή τη Επιτροπή Έμβηση εκείνη τη συνεδρίαση. Λοιπόν, το πρώτο καλό νέο από αυτή την αξιολόγηση είναι ότι το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο έχει φέρει αποτελέσματα δεν έχει υπάρξει κάποια σημαντική ε, κρίση ε, μετάδοση ασθένεια από την υιοθέτηση των ε, νομοθετημάτων αυτών και μετά. Έτσι, ο ιός του Δυτικού Νείλου, για παράδειγμα, περιορίστηκε, παρεμποδίστηκε. Και τα δεδομένα που έχουμε για τις σοβαρέ παρενέργειες, οι αντιδράσεις μας δείχνουν μόνο μία στις χίλιες μονάδες. Και αυτό είναι εξαιρετικό αποτέλεσμα και οι περισσότεροι από όσου απάντησαν στη διαβούλευση είπαν ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά την άποψή του αύξησε την ασφάλεια και την ποιότητα και αυτό δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί τόσο καλά μόνο σε εθνικό επίπεδο. Πάμε και σε κάποιες ανησυχίες που προκύπτουν από την αξιολόγηση οι ανησυχίε αυτέ σχετίζονται κυρίω με το κατά πόσο τα πλαίσια θα μπορούν να έχουν εφαρμογή στο μέλλον. Πέντε καραντίνες ε, εμφανίζονται ε, με κάποιο ιδιαίτερο χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα κάποιε τεχνικέ διατάξει φαίνονται απερχαιωμένε. διότι οι τομεί του αλλάζουν ταχαίως, διαρκείς τεχνολογικές εξελίξεις, νέοι κίνδυνοι, όπω είπα, κοινωνικέ αλλαγέ επίση, Από την άλλη, οι νομοθεσία συχνά είναι ιδιαίτερα λεπτομερεί και είναι δύσκολο να την αλλάξει κανεί έγκαιρα. Και επίση η νομοθεσία δεν καλύπτει νέε θεραπείε όπω τη χρήση μητρικού γάλακτο ή ε, κάποιε άλλε ε, μεταμοσχεύσεις. Ε, το δεύτερο που είδαμε ότι είναι, αυτές οι διατάξεις δεν μπορούν να, εφαρμοστούν εύκολα στις μεταγγίσεις πλάσματος και κυτάρων. Είναι ταχύως ε, εξελισσόμενοι τομεί αυτοί, οπότε απαιτούν να αυξήσουν τα σχετικά μέσα και τις ικανότητες και οι εθνικές ε, αρχές. Ε, η τωρινή συχνότητα των διετών ελέγχων φαίνεται να μην επαρκεί και φαίνεται να μην είναι αρκετά διαφανεί κάποιε διατάξει. Κάτι τρίτο που διαπιστώθηκε είναι ότι κάποιοι πολίτε μπορεί να μην προστατεύονται παρκώ. Απαιτούνται όλο και περισσότεροι δωρητέ λόγω τη αυξανόμενη ζήτηση ή των αναγκών ή του εμπορικού ενδιαφέροντο. Ωστόσο, είναι περιορισμένε οι διατάξει που προστατεύουν το follow-up των δωρητών. Και επίση λοιπόν διατάξει για την καταχώρηση και την παρακολούθηση τη υγεία των παιδιών που γεννιόνται από το IVF. Ε, μακροχρόνια Επίσης βρεθήκαν κάποια προβλήματα στην καινοτομία. Δεν διευκολύνεται η καινοτομία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι καινοτόμε θεραπείες απαιτούν καινοτόμε διοδοτήσει, συμπεριλαμβανομένη τη αποτελεσματικότητας έγκρισης. Αυτό είναι όλο και πιο δύσκολο η περιπλοκότητα και λόγω της περιπλοκότητας και των προόδων αυτού του τομέα. Πράγματι, πολλές καινοτομίες ε, ε, ε επικαλύπτουν ε, πολλά νομικά πλαίσια ε, και έτσι χρειάζεται περισσότερη σαφήνεια. Το άλλο τελικό βασικό πόρισμα είναι ότι είναι περιορισμένες οι διατάξεις ε, διασφάλισης της επάρκειας. Βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό στη ΣΥΠΑ για το πλάσμα και για κάποια διεστών. Επίσης, όσον αφορά την ε, ετοιμότητα για έκτακτες ανάγκες, αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωση των μέτρων. Περισσότερες λεπτομέρειες φυσικά μπορείτε να βρείτε εδώ όλη την αξιολόγηση σε αυτή την εδώ τη διεύθυνση που βλέπετε εδώ. Αλλά ουσιαστικά αυτά ήταν τα κύρια απορίσματα της αξιολόγησης για το αίμα, τους ιστούς και τα κύτταρα. Η Κομισιόν φυσικά σημειώνει πολύ προσεκτικά όλα αυτά μαζί με άλλα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διαθεσή μου όπως τις ανησυχίες που έχουμε διαπιστώσει που προέκυψαν κατά τις διαβουλεύσεις αλλά και το παρόν κοινοβούλιο που ζητά ενισχυμένη συλλογή του πλάσματο όπω υιοθετήθηκε σε ένα κείμενο στι αρχέ του έτου. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά και θα μα βοηθήσουν να χαράξουμε το επόμενο βήμα ε, που θα είναι η αποφάση της Κομισιόν ε, λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, εμπεριστατωμένη παρουσίαση. Ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνη <coughs> πολλές φορές το σύστημα. Πριν δώσω το λόγο συναδέλφους, δεν ξέρω αν έχουμε εκπροσώπους από το κόμμα. Κυρία Λάγκε, θέση του κυρίου Λάγκε. Αυτή η παρουσίαση της Επιτροπής δείχνει ποιες δυσκολίες υπάρχουν. Διότι βασικά είπατε ότι η νομοθεσία ήθελε να εξασφαλίσει την ε, ασφάλεια των ε, συστατικών αυτών. Και βεβαίως υπάρχει και θέμα ηθικής, υπάρχουν νέες υπηρεσίες, η διαθεσιμότητα τέτοιων ουσιών βεβαίως έχει να κάνει και με θέματα ηθικής και με θέματα εθνικής νομοθεσίας και θα ήθελα να μου πει η Επιτροπή πώς πιστεύει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε δεδομένου ότι τα θέματα ασφαλείας ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση ξεπερνιόνται από τα θέματα ηθικής καμιά φορά. Επίσης, το θέμα της διασυνοριακής ε, συνεργασίας σε τέτοιου περιπτώσεις. Τι γίνεται. Τέτοιε λοιπόν αίμα, ιστός, κύτταρα ε, μεταφέρονται διασυνοριακά. Επίσης, τι γίνεται με την ε, νομοθεσία που ισχύει σε μια χώρα αλλά δεν ισχύει στην άλλη. Άρα δυσκολεύει όλη αυτή η συνεργασία. Τι γίνεται λοιπόν δεν συνοριακά. Και επίσης, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με την ε, νομοθεσία για τα, για την, για τα οάρια, θα πρέπει να υπάρχει πλήρη συγκατάθεση. Στην Ισπανία, Φερρυπίν, για να δωρήσετε ο Άρια, ε, πληρώνεστε. Σε άλλες χώρες όχι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό σε ε, θελούσια βάση χωρίς να υφίσταται κανείς ε, πίεση για να δωρήσει. Τι προβλέπει η νομοθεσία. Ο κύριος Νικόλας Γκονσάλες αρίές από το ΕΣΕΝΤ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτά τα οποία μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και έχουμε την ε, σχετική οδηγία συμφωνούν ναι, με αυτά τα οποία όλους μας απασχολούν. Όχι μόνο η βιοασφάλεια, η ύπαρξη νέων ασθενειών από άτομα τα οποία ίσως έρχονται από άλλες υπήρους. Τα θέματα των ελέγχων ε, του αίματος, των κυτάρων, των ιστών πρέπει να είναι πάρα πολύ αυστηρός. Για λόγους ηθικής επίσης κάτι αναφέρθηκε. Ξέρουμε ότι χρησιμοποιούνται δωρητές, δωρήτριες μάλλον, μητρικού γάλακτος και το γάλα αυτό, από τις μητέρες αυτές, αποστέλλεται ως εμπορικό προϊόν σε μωρά που έχουν γεννηθεί πρόοδα, πρόωρα για να υποκαταστήσει το γάλα που πρέπει να πάρουν. Ας το ξαναεξηγήσω μάλλον πιο απλά μέσω οργανώσεων ε, που δεν έχουν οικονομικά συμφέροντα, συλλέγεται μητρικό γάλα, το γάλα αυτό ξηραίνεται και επειδή δεν μπορεί να πολιθεί ως μητρικό γάλα στην κανονική αγορά, γίνεται προσπάθεια να πολιθεί για τα πρόωρα μωρά στα νοσοκομεία. Διότι η μητέρα ίσως δεν μπορεί να θυλάσει το πρόωρο μωρό της. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, το έχετε αντιμετωπίσει, μπορείτε να το συμπεριλάβετε στη νέα οδηγία. Και τελικά, αυτό το οποίο είπατε για τα οάρια, ε, συνάδελφε, στην Ισπανία. Ξέρω ότι και σε άλλες χώρες πληρώνονται αυτού του είδους οι δωρεές. Πώς μπορεί κάτι τέτοιο να το ρυθμίσει με κανονισμούς και το, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, όλοι εμείς. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Διαπτορινιό Τχιγέγλου Ενουάρ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δεδομένου ότι είμαστε λίγοι, επιτρέψτε μου και εμένα να υποβάλω στον κύριο Γενικό, στον Απρίλιο, το Γενικό Διευθυντή, πολλές ερωτήσεις, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πολύ σαφή παρέμβασή του, που μας ενημέρωσε πάρα πολύ για το όλο θέμα. Όσον αφορά το πλάσμα, ξέρουμε ότι πολλοί ασθενείς που έχουν ε, ε, ε νοσήματα ή άλλου είδους νοσήματα χρειάζονται πλάσμα. Αυτό είναι και θέμα δημόσιας υγείας. Είπατε επίσης ότι εξελίσσεται η νομοθεσία και αποκαλύπτει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται από την εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων τέτοιων στατικών που έρχονται κυρίως από τη ΣΥΠΑ. Κάτι τέτοιο μπορεί να δημιουργήσει πλήρη εξάρτηση ε, όσον αφορά την προσφορά. Άρα θα πρέπει να λάβουμε μέρος ώστε να έχουμε τα κατάλληλα αποθέματα. Επίσης αναφέρθηκε το θέμα του διαφορετικού τρόπου ευχαριστίας των δωρητών. Εγώ είμαι από τη Γαλλία, που είναι μια χώρα η οποία προσδίδει μεγάλη σημασία στην εθελούσια ε, δωρεά για ηθικούς και για άλλους λόγους. Καταλαβαίνω ότι άλλα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικά πρότυπα. Τι μέτρα προβλέπετε να ληφθούν ώστε να μπορέσει να συλλέξει η Ευρωπαϊκή Ένωση μεγαλύτερες ποσότητες πλάσματος, να γίνει πιο ανεξάρτητη από τη ΣΥΠΑ και βεβαίως να ε, το κάνει αυτό σεβόμενοι και τα δύο συστήματα, πράγμα απαραίτητο. Επίσης υπενθυμίσατε ότι η συνέχεια της προσφοράς απειλείται και τις κλιματικές αλλαγές και από το γεγονός ότι έχουν φτάσει και στην Ευρώπη κουνούπια που μεταδίδουν την τσίκα ή την τσικουγκουνιά ως ασθένειες. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Στη δική μου την πόλη έχω ένα τέτοιο παράδειγμα που η αιμοδοσία πρέπει να πω ότι σταμάτησε δεδομένου ότι παρουσιάστηκαν τέτοιου είδους τροπικές ασθένειες, άρα η αιμοδοσία δεν μπορούσε να γίνει. Για να κάνουμε μια διασύνδεση με το θέμα που εξετάσαμε προηγουμένως, με τη θέματα της πολιτικής προστασίας, τι πέτρα προβλέπετε να πάρετε, ώστε να μπορέσετε να αμβλύνετε τους κινδύνους που υπάρχουν σε περίπτωση ε, κρίσης σε θέματα υγείας. Σήμερα το πρωί μου υπενθύμησε κάτι μια οικογένεια ασθενούς μου. Υπάρχει θέμα κατανομής των, ε, δε, των, ε, των βλαστοκυτάρων, των περιφερειακών και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ε, διαφοροποίηση μεταξύ των ε, δωρητών μυελού των οστών για να θεραπευτούν σε κάποιες χώρες άλλες εκτός της δικής μου τέτοιες σοβαρές ασθένειες ε, πώς μπορείτε τέτοιους ανημιογένειες να τις αμβλύνετε. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω εδώ παρόντες τους συντονιστές. Δεν βλέπω να είναι εδώ οι συντονιστές, οπότε θα πάρει το λόγο ποιος το επιθυμεί. Παρακαλώ κύριε Στέφαν Γιούτε, Σας ευχαριστώ πρόεδρε και σας ευχαριστώ επειδή καλωσορίσατε το μελλοντικό, τους μελλοντικούς μας συμβούλους που είμαι ευτυχής που είναι σήμερα εδώ ε, για μια πολύ σημαντική ε, συνεδρίαση. Θα τα πω τώρα ρουμανικά ε, για ευνόητους λόγους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, θέλω να πω ότι στην ακρόαση της Τέλης ε, Κυριακίδη συζητήσαμε για όλα τα προβλήματα που έχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα Υγείας ε, γιατί υπάρχουν πολλοί περιορισμοί. Ταυτόχρονα όμως ο Ευρωπαίος πολίτης δεν το γνωρίζει και έχει μεγάλες προσδοκίες. στη χώρα μου, τη Ρουμανία, θα πρέπει να σας πω ότι τα προβλήματα υγείας είναι μεταξύ των top 5 των ανησυχιών των πολιτών. Ο πολίτης δεν καταλαβαίνει αυτά τα λεπτά ζητήματα της αρμοδιότητας και της στήριξης. Ξέρει μόνο πως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να βοηθήσει. Όπως έλεγε λοιπόν και η συνάδελφος Τριγέλε ε, υπάρχουν ε, περιστάσεις επίγουσας ε, ανάγκης. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας στη χώρα μου ήδη το 2018 είχε υποβάλει αίτημα για θέματα υγείας επειδή δεν υπήρχαν δεν υπήρχαν αποθέματα αιμοσφαιρίνης γιατί αν θυμάστε έχει υπάρξει ένα ατύχημα στο Βουκουρέστι σε μια δισκοτέκ όπου υπήρξαν πολύ τραυματισμένοι, χρειαστήκαμε ιστούς, αίμα, πλάσμα. Ρωτώ λοιπόν ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τα όσα μπορεί να νομίζει ο πολίτης αλλά και τις πραγματικές ανάγκες του πολίτη. Εγώ θα παρακολουθήσω πολύ, πολύ εκ του συναγκής τα όσα συμβαίνουν όχι μόνο σε ε, επίπεδο μηχανισμού πολιτικής προστασίας αλλά και για θέματα υγείας όπως αυτό που μας απασχολεί τώρα. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω κάποιος άλλο να ζητά το λόγο, οπότε θα δώσω το λόγο στον, ε, κύριο, στον αρμόδιο να απαντήσει στα σχόλια των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Είναι αλήθεια ότι διάφορα ζητήματα περιλαμβάνουν πτυχή ασφάλειας αλλά και ε, ηθικές, ηθικής δεοντολογίας. Όπως είπαμε, αυτή η νομοθεσία ασχολείται με την ε, ποιότητα και την ασφάλεια και ο χειρισμός συνολικός αυτών των θεμάτων θα απαιτήσει συνδυασμό μέτρων. Μέτρων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και υποστηρικτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν σε εθνικό επίπεδο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα προβληματιστεί η Επιτροπή και θα το λάβει υπόψη. Ετέθη το ζήτημα της διασυνοριακής πτυχής. Πράγματι, αυτό αυτό το θέμα ήταν αυτό που πυροδότησε την ε, νομοθεσία αυτή. Είναι μια σημαντική πτυχή και ε, διάφορες απαντήσεις μπορούν να δοθούν. Καταρχάς, ε, γι' αυτό έχουμε κοινούς κανόνες ώστε να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον εντός της Ένωσης θα ισχύουν τα ίδια στάνταρ ποιότητας και ασφάλειας. Ωστόσο, αυτό οδηγεί στη δεύτερη παρατήρηση που έγινε για την αξιολόγηση. Αν τα... και κατά πόσο τα κράτη-μέλη έχουν διαρκείς ε, δυνατότητες για να εφαρμόσουν τους κοινούς κανόνες. Ε, πολλές φορές υπάρχουν σημαντικές διαφορές ε, στις δυνατότητες των κρατών μελών και εκεί χρειάζεται περισσότερη δουλειά. Να θυμίσω ότι δουλεύουμε χέρι με χέρι με το Συμβούλιο τη Ευρώπης που έχει κάνει εκτεταμένο έργο για αυτό το θέμα, όπως α πούμε και για την ιδεοντολογία. Και βεβαίως το Συμβούλιο της Ευρώπης εκτελεί και δικές του μελέτες ας πούμε, σε σχέση με αυτό που ρώτησε ο, ο κύριος Ευρωβουλευτής για τις στατιστικές, το Συμβούλιο ασχολείται πολύ, γιατί είναι κινούμενη η, εικόνα. Γνωρίζουμε όμως ε, αρκετά καλά ότι υπάρχει μεγάλη διασυνοριακή κίνηση ιστών και κυτάρικων ιστών. Για το θέμα της εθελοντικής δωρεάς ε, αίματος, πλάσματος ε, κτλ. Το θέμα της εθελοντικής δωρεάς είναι μια ισχυρή σύσταση μέσα στο πλαίσιο του νομικού, το μας και όλα τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει αυτή την αρχή, αν και η εφαρμογή διαφέρει λόγω τη τοπική πραγματικότητα. Υπάρχουν, όπω αναφέρατε, διαφορετικέ εθνικέ προσεγγίσεις που είναι επίση κατανοητέ, διότι η κατάσταση διαφέρει όντω από χώρα σε χώρα και επίση ε, κάποιες χώρες έχουν ε, ε, διαφορετικές απαιτήσεις. Η αξιολόγηση της ε, αιμοδοσίας προέκυψε, μας έδωσε μάλλον στοιχεία σε σχέση με την προστασία των δοτών και σε σχέση με τα πρότυπα που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες. Για όλα τα πρότυπα, όλα τα μοντέλα υπάρχει ισχυρή απέτηση για την ενίσχυση της προστασίας των δεδομένων των δοτών εκεί όπου χρειάζεται να αυξηθεί η ε, η αιμοδοσία είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν και να εφαρμόζονται μέτρα προστασίας των πληροφοριών περί δοτών. Είναι ένα μέτρο λοιπόν που θα πρέπει να ισχύσει σε όλα τα κρατημέλη άσχετα με την προσέγγιση που έχουν. Τώρα, για το συγκεκριμένο θέμα του ανθρώπινου μητρικού γάλακτος. Είναι ένας τομέας που δεν καλύπτεται από την νομοθεσία και η αξιολόγηση αυτή το έδειξε ότι δηλαδή θα πρέπει αυτό να το διερευνήσουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η νομοθεσία θα εξυγχρονιστεί και θα ακολουθήσει τις ε, σύγχρονες ε, εξελίξεις. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες είναι πιο πρόσφατες λοιπόν. Για το θέμα της ζήτησης πλάσματος. Καταρχάς το πλάσμα είναι σημαντικό αφ' αυτού. Είναι είναι ένα πολύ σημαντικό ιατρικό προϊόν, το οποίο όλο ένα και περισσότερο είναι το σημείο κίνησης για διαφόρων ειδών θεραπευτικά προϊόντα. Είναι σαφές ότι στην Ευρώπη έχουμε μια κατάσταση γενικής εξάρτησης. Περίπου το μισό του ανάγκη μα σε πλάσμα προέρχεται από τη ΣΥΠΑ. Είμαστε πολύ πίσω δηλαδή από την ε, αυτάρκεια. Και αυτό θα το έλεγα ανεξάρτητα από τα συστήματα των κρατών μελών. Δεν υπάρχει κανένα κρατός μέλος που να έχει επιτύχει αυτάρκεια σε αυτό το θέμα. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Καταρχάς να ενισχύσουμε την προστασία των δοτών, να, δώσουμε, να, κινητοποιήσουμε την δωρεά αίματος και πλάσματος, δηλαδή οι πολίτες δεν γνωρίζουν ότι μπορούν να δώσουν και πλάσμα, περισσότερο ξέρουν ότι μπορούν να δώσουν αίμα, αλλά για πλάσμα δεν ξέρουν πολλοί πολίτες. Και επίσης ε, θα έχουν υπάρξει σημαντικές τεχνολογικές και επιστημονικές πρόοδοι που εξασφαλίζουν τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε πλάσμα για την εξαγωγή δηλαδή συγκεκριμένων προϊόντων από το πλάσμα, ώστε να μπορούν περισσότεροι αποδέκτες να ωφεληθούν από τα συστατικά του πλάσματος, να γίνει δηλαδή ευρύτερη χρήση του πλάσματος που πράγματι συλλέγεται. Μία από τις πιο σημαντικές απειλές που έχουμε είναι η απειλή από νέες ασθένειες, νόσους, παθογόνες που μπορεί να οφείλονται ε, ίσως στη ρήπανση, ίσως στις κλιματικές αλλαγές. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε αυτάρκεις, γιατί η γεωγραφική, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης είμαστε εκθεθειμένοι. Ε, μάλλον οι ΙΠΑ είναι πιο ο, Η ΙΠΑ ε, εκτίθεται, ας πούμε στο ΖΙΚΑ για παράδειγμα λόγω της γεωγραφικής του θέσης, ενώ εμείς όχι. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε πιο αφτάρκες η ευρωπαϊκή πρόληψη και έλεγχο έχουν επίση βελτιώσει τι δραστηριότητέ του εποπτεία ώστε να εξασφαλίσουμε πω παρακολουθούμε στενά τι γίνεται και να είμαστε σε θέση να προλάβουμε αυτού του κινδύνου. Και έπειτα υπάρχουν και τεχνολογικέ και επιστημονικέ εξελίξει για να εξασφαλίσουμε την ποιότητα του πλάσματο μέσω διαφόρων τεχνολογικών ελέγχων, όπω α πούμε αφαίρεση αυτών των παθογόνων και των ιών από το πλάσμα και το αίμα που συλλέγονται. Τέλος, όσον αφορά τις διαφορές στα στοιχεία. Ναι, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στα στοιχεία. Αυτό συνδέεται και με τις ικανότητες των 100 μελών. Γιατί βέβαια αυτό σημαίνει πως οι χώρες που έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν τα στοιχεία με αξιόπιστο τρόπο ε, για να έχουν πλήρη έλεγχο της κατάστασης είναι λιγότερο. Και εδώ πρέπει να προσέχουμε πολύ, να δούμε ποια είναι τα πορίσματα αυτής της αξιολόγησης, πώς μπορούμε να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη για να αυξήσουν τις δυνατότητές τους με διάφορους τρόπους και σας ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα χρησιμοποιήσω το ιδιότητά μου ως Προέδρου για να σας ρωτήσω μια ερώτηση που ξέχασα προηγουμένως να υποβάλω. Κάτι που συζητάμε εδώ είναι εάν θα πρέπει να κάνουμε έκθεση πρωτοβουλία για αυτό το θέμα και αν υπάρχουν νομοθετικέ προτάσεις που θα έρθουν από την Κομισιόν σχετικά με αυτά που θέλουμε. Αυτό θα μας ε, ε, δώσει μια εικόνα. Έχετε εσεί υπόψη κάποιο χρονοδιάγραμμα για την αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας. Είστε σε θέση να με ενημερώσετε για το ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τη Κομισιόν. Βέβαια, Έχοντα υπόψη πάντα πω μόλι ανέλαβαν νέοι επίτροποι. Ναι, βεβαίω, όπω ξέρετε, μόλι τριών χρονών είναι, η, τριών ημερών είναι μάλλον η καινούργια επιτροπή. Όπως σας είπα, έχουμε πολύτιμα στοιχεία που θα υποβάλουμε ε, για να ληφθούν αποφάσεις. Έχουμε πολλές πληροφορίες ε, που, στις οποίες μπορούν να βασιστούν οι σχετικές αποφάσεις και αυτό βεβαίως σχετίζεται και με άλλες προτεραιότητες ε, που είναι στην ατζέντα της Κομισιόν, όπως ας πούμε το θέμα της παροχής βασικών φαρμάκων, που όπως ξέρετε περιλαμβάνεται στην αποστολή του χαρτοφυλακίου της Επιτρόπου κυριακή Και βέβαια το πλάσμα, κύτταρα, ιστή είναι όλο ένα και περισσότερο υλικά για ε, πολύ προηγμένες θεραπείες αλλά και προηγμένα φάρμακα. Ε, βεβαίως πρώτο βήμα θα είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ασφαλή ε, προμήθεια, ε, ποσότητα αλλά και ποιότητα και ασφάλεια. Είναι πολύ σημαντικό γιατί όπως σας είπα είναι και υλικό, πρώτη ύλη για την ε, παραγωγή άλλων θεραπευτικών ε, ε, φαρμάκων ή και θεραπείων. Η Κομισιόν πολύ σοβαρά λοιπόν θα πρέπει αυτό να το λάβει υπόψη και έχουμε πολύ καλά στοιχεία από τον οποίων να βασίσουμε συστάσεις και ενδεχομένως λήψη αποφάσεων. Ευχαριστώ. Ακούγονται πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά. Θα περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι πολιτικές αποφάσεις. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα για να σας ενημερώσω. Α, δεν υπάρχουν περαιτέρω ανακοινώσει εδώ. Σα ευχαριστώ για τις εισηγήσει Μάλιστα. Έχετε τίποτα άλλο να πείτε στα διάφορα τώρα. Γιατί αν όχι, ε, να σας ενημερώσω ότι η επόμενη συνεδρίαση τη Επιτροπής μας θα γίνει στις 16 Δεκεμβρίου. Περιμένουμε να έχουμε έκτακτη συνεδρίαση στο Στρασβούργο στις 16 και μετά η επόμενη συνεδρίαση μπορεί να είναι στις 9 Ιανουαρίου 2020, δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι, μπορεί αυτό να ακυρωθεί, αλλά αυτοί, αυτές προσωρινά είναι οι ημερομηνίες. μεγάλη μέρα είχαμε σήμερα, αρχίσαμε στις 9.30 το πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ όσοι σας αντέξατε όλη την ημέρα, ευχαριστούμε που ήρθατε, ευχαριστώ τους επισκέπτες. Ελπίζουμε να μάθατε κάποια πράγματα. Ευχαριστώ την γραμματεία και τους διερμηνείς. Ε, σταματάμε λίγο νωρίτερα, πράγμα που είναι πάντοτε ευχάριστο.